A ver, un poco de orden. Λοιπόν, λίγο ησυχία παρακαλώ. Καθίστε παρακαλώ, αργήσαμε πρέπει να ξεκινήσουμε. Please. Καπόουλας, Madame Ροδούς. Παρακαλώ καθίστε κύριε Ρότχα, κυρία κύριε Καπούλας. Καλημέρα σε όλους να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλίας. Έχετε την ημερήσια διάταξη. Σας παρακαλώ λίγο ησυχία. Κύριε Κούν, παρακαλώ. Μίστερ Κούν. Estamos, eh, vamos a aprobar el orden del día. Να εγκρίνουμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη. Εάν δεν έχετε πρόβλημα, θα ήθελα να σας ενημερώσω για δύο αλλαγές που θα γίνουν. Καταρχάς, το σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης, πρόταση για τα τεχνικά μέτρα της Βαλτικής θα είναι το σημείο 19α και το σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης, που είναι μία από τις εκθέσεις του κυρίου Γκάλαγκερ, θα είναι το 7ο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Εάν συμφωνείτε λοιπόν με αυτές τις τροποποιήσεις και δεν έχετε κάποια άλλη να προτείνετε, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Επίσης να σας πω ότι δεν υπάρχει διερμηνία από τα σουηδικά. Η κυρία Λεβίν το ξέρει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο ο οποίο ακούει σουηδικά. Υπήρξαν κάποια προβλήματα και δεν υπάρχει σουηδική καμπίνα σήμερα. Επίση, να σα ε, ενημερώσω ότι ω συνήθω η συνεδρία μεταδίδεται μέσω του Europal TV να εγκρίνουμε τώρα τα πρακτικά της 1ης και 2ης Ιουνίου. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις στη διάρκεια των δύο ημερών της συνεδρίασης της Επιτροπής Αλίας, θα θεωρούμε ότι έχουν εγκριθεί. Τέταρτον, ανακοινώσεις της Προέδρου. Προς το παρόν δεν έχω τίποτα να σας ε, πω. Να περάσουμε λοιπόν απευθεία στην ψήφιση της έκθεσης της ονομοδότησης συγγνώμη, του κ. Εντινόρου για την ε, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Ε, ελπίζω να έχετε όλες τις κάρτες ψηφοφορίας για να ψηφίσουμε. Ο κύριος Αντινόρα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα δύο λεπτάκια να ευχαριστήσω τη Γραμματεία, κυρίως τον κύριο Χιμένες, διότι μας προσέφερε ουσιαστική βοήθεια να ευχαριστήσω επίσης όλους τους κοιόδης εισηγητές για την έκθεση και ε, τους βοηθούς και όλους όσους μας επέτρεψαν να έχουμε την γνωμοδότηση που έχουμε. Θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι η πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η συνθήκη της Λισαβόνας που εμείς ως Επιτροπή Αλίας ε, χρησιμοποιούμε τη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, οπότε σήμερα ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που ε, χρησιμοποιούμε τους κανόνες ε, που ναι μεν είναι ήδη ενισχύει, αλλά που θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε και τα επόμενα χρόνια. Ε, γνωρίζετε όλοι νομίζω πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ Επιτροπής Αλλιές και Επιτροπής Μεταφορών και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Πρόεδρο Φράγκα διότι ξέρετε ότι η μάχη είναι εν εξελίξη για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα και θα ήθελα να εξηγήσω, διότι με κάποιου μιλήσαμε με ένα, αλλά ίσω δεν δόθηκε δυνατότητα να μιλήσω με όλου του συναδέλφου, ότι εάν υπήρξαν αμφιβολίες σε κάποιες ε, τροπολογίες και Είχαμε, αν όχι απαραίτητα αρνητική άποψη, ζητήσαμε όμως απόσυρση, τροποποίηση σε κάποιες περιπτώσεις ή ε, ήμασταν αντίθετοι στις... Ε, συμβαστικέ λύσει που τώρα συμπεριλαμβάνονται στην ε, γνωμοδότηση ήταν γιατί εμεί, ω Επιτροπή αλληλία, μπορούμε να επισέλθουμε στα θέματα αυτά μόνο σε όσα άπτονται τι αρμοδιότητές μα. Ορισμένε φορέ είχαμε κάποιε τροπολογίε οι οποίε υπερεύαιναν τι αρμοδιότητε τη επιτροπή αλληλία και μπαίναμε σε διαφορετικέ αρμοδιότητε, παραδείγματο χάρη μεταφορέ, περιβάλλον, αρμοδιότητε άλλων επιτροπών. Αυτό δεν επιτρέπεται βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα και ίσω να μας έφερνε και ενώπιον μιας κατάστασης ε, στην οποία η Επιτροπή Μεταφορών θα έλεγε όχι ε, και μάλιστα δικαιολογημένα γιατί θα είχε και τον κανονισμό που θα την κάλεπτε. Εάν λοιπόν ε, κάποιες στιγμές διαφωνίας, ε, αν θέλετε, ή διαλόγου προέκυψαν ήταν ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ε, κατά τα άλλα θεωρώ ότι καταλήξαμε σε μια καλή συμβιβαστική συνολική πρόταση. Υπήρχαν και επιμέρους συμβιβασμοί, αλλά ελπίζω ε, στη συνέχεια με την Επιτροπή Μεταφορών να μην έχουμε πρόβλημα, να σεβαστεί τη γνωμοδότησή μας και να καταλήξουμε τελικώς στην Ολομέλεια και να εγκριθεί το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Gracias. Bueno, pues empezamos el, el voto, entonces. Ωραία, να ψηφίσουμε. Συμβαστική πρόταση 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογίε 1, 2, η τρία είναι συμβατή, όχι, καταπίπτει και αυτή. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 4 του κυρίου ε, Φερέιρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5, κυρία Πατράου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 10 υπέρ, 10 κατά, καταπίπτει. Η 6 αποσύρεται, συμβιβαστική πρόταση 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 7, οι 8, συμβιβαστική πρόταση 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 9, οι 10 και ψηφίζουμε την τροπολογία 11 της κυρίας Ιώτοβα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 12, 13, 15 και ψηφίζουμε την τροπολογία 16 του κ. Φρέιρα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18, Πατράων Νέβες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Ρέιμερς Χάγκλουντ Γένσεν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Ρόντος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 του κυρίου Φερέιρα. Άρχεται η ψηφοφορία. ...πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24 του κυρίου Κάντεκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 του κυρίου Αρσένη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 του κ. Αρσένη, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογ... Συμβιβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 27, 28 και ψηφίζουμε την τροπολογία 29 του κ. Φερέιρα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30 Πατράων Νέβας. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31 της κυρίας Πατράου Νέβες, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32 αποσύρθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 33 και 34. Ψηφίσουμε την τροπολογία 35 του κυρίου Τσουκουρλά κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα, που είναι το υπόλοιπο κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 10 υπέρ 10 κατά καταπίπτει. Η 36 αποσύρεται και η 37. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 8, να το ψηφίσουμε τώρα, άρχεται η ψηφοφορία. Σε Πέραση τη ψηφοφορία. Υπάρχουν κάποιοι που δεν ψήφισαν. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 αποσύρεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 38 και οι 41. Τροπολογία 39 του κυρίου Αρσένη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40 του κυρίου Αρσένη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42 του κ. Αρσένη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 44 αποσύρεται. Η τροπολογία 45 Τη 45. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46 αποσύρεται. Η 43 ψηφίστηκε και απορρίφθηκε, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, να ψηφίσουμε τη 43. Έχετε δίκιο, δεν την ψηφίσαμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Εντάξει, ψηφίσατε. Μην ανησυχείτε. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 47, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα της τροπολογίας 47, άρχεται η ψηφοφορία. Σε η la votación, Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Καταπίπτει. Συγγνώμη, απορρίπτεται. Τροπολογία 23 του κυρίου Φερέιρα. συγγνώμη, η 23 καταπίπτει, επομένως ψηφίζουμε τη 48 της Πατράων Νέβες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε λοιπόν τώρα τη γνωμοδότηση ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. 19 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 1 αποχή εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Τινόρο. Και με αυτό ολοκληρώθηκε το σημείο υπαριθμών 6 και περνάμε, συγγνώμη, 5 και περνάμε στο σημείο 6. Θα το δούμε μαζί με το σημείο 7 της ημερησίας ε, τα τα πολιετή για ε, το Σαφρίδι και για το γάβρο στο φυσικαϊκό κόλπο, όπως ε, θα θυμάστε, σε αυτές τις δύο εκθέσεις. Οι δύο αυτές εκθέσεις εκπονήθηκαν. Σας παρακαλώ, λίγη ησυχία λέει η Πρόεδρος, γιατί δεν μπορώ να μιλάω με τόσο θόρυβο. Οι δύο εκθέσεις λοιπόν εκπονήθηκαν πριν τη σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα. και αφού τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα, υλοποιήσαμε μία ψηφοφορία πρώτων συναντηλισμού έτσι ώστε οι συγητές να μπορούν να διαπραγματευτούν με το Συμβούλιο για να μπορέσουν να φτάσουν σε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Αυτό ήταν ο στόχο. Όπω ξέρετε, αυτοί οι φάκελοι έχουν παραλύσει καθώ το Συμβούλιο τόσο για τον Γαβρού και για το Σαφρίδη έχει αλλάξει την ε, νομική βάση και υπάρχει μία γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου για το θέμα του Σεφριδίου, η οποία είναι υποεκπώνηση. Και αυτή η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου δικαίωσε τη θέση του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, η νομική βάση κατά αυτού θα έπρεπε να είναι το 43-2 και όχι το 43-3 που είναι αυτό που ζητά το Συμβούλιο. Και έτσι λοιπόν, για να σας πω τι σημαίνει το 43-3 ότι θα καταργούσαν τη συναπόφαση. Για μας λοιπόν αυτό θέμα είναι κάσους Για την περίπτωση του Γαύρου δεν υπάρχει ακόμη γνωμοδότηση, αλλά ελπίζουμε να υπάρχει. Δεν σημαίνει όμως ότι το Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει την ε, άποψη της νομικής υπηρεσία του με μία ε, νομική γνωμοδότηση. Είναι δύο νομικές γνωμοδοτήσεις που υποστηρίζουν ε, την θέση του Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά το Συμβούλιο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αν εγκρίνουν το 43-3, τότε νομίζω ότι θα έπρεπε να προσφύγουμε στο 10, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί στο μέλλον αυτό θα σημαίνει ότι όλα τα πολιετή σχέδια θα μπορούσαν να περάσουν στα χέρια του Συμβουλίου και να καταργηθεί η τακτική νομοθετική διαδικασία, η συναπόφαση δηλαδή. Έτσι λοιπόν, να δώσω το λόγο τώρα στους δύο συγητές για να μας πούν ποια είναι η θέση τους και πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε στην περίπτωσή τους. Και στη συνέχεια θα ανοίξουμε και το βήμα. Θα κάνουμε μία συζήτηση έτσι λοιπόν. Έτσι όπως έχουμε εδώ τη σειρά στη μισή διάταξη, καταρχήν ο κύριος Γκάλεχερ και κατόπιν η κυρία Μπιλμπάου. Παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που παρουσιάσετε αυτή την εισαγωγή στις εκθέσεις αυτές ε, όπου είμαι εισηγητής εν ονόματι αυτής της Επιτροπής για να παρουσιάσω την ε, κατάσταση ε, η οποία διαμορφώθηκε και μάλλον το σπηλίστηκε από την ε, είσοδο σε εφαρμογή της συνθήκης της ε, Λισαβόνας έγινε μία πρώτη ψηφοφορία τον Δεκέμβριο που διατύπωσε την άποψη του Κοινοβουλίου και έκτοτε συναντήθηκα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και είχα την εντύπωση ότι είχαμε προχωρήσει πολύ. Μέχρι ότου συναντήθηκα με την κυρία Δαμανάκη για να ακούσω ότι η δικιά μου εντύπωση ήταν αθασμένη και απέσυρε την ανακοίνωση αυτή ενώ είχε ε, συστήσει να τροποποιηθεί. Είχαμε συναντηθεί με την ε, Επιτροπή και με την Επίτροπο και είχε πει σαφώς ότι ήταν υπέρ του να τροποποιήσει ε, το κείμενο. Κατόπιν αυτού όμως άλλαξε γνώμη και επέτρεψε να προχωρήσει το θέμα υπό έναν όρο ότι δεν θα αποτελέσει προηγούμενο για επερχόμενες εκθέσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι το Συμβούλιο είχε λάβει νομική συμβουλή ότι πρέπει να βασιστεί στο άρθρο 43.2 το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης και στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο πίστευε ότι έπρεπε να βασιστεί στους 43-3 οπότε το Συμβούλιο είχε αποκλειστική εξουσία. Άρα εμείς πρέπει να επιμείνουμε διότι αν επιτρέψουμε αυτό να προχωρήσει βάση του 43-3 τότε θα εξυπηρετήσουμε δυσμενώς όχι μόνο το Κοινοβούλιο αλλά θα δημιουργήσουμε και ένα προηγούμενο Οπότε σχετικά με την άλλη έκθεση νομίζω ότι ε, σωστά ε, βασιστήκαμε στο 43-2. Θέλαμε ε, να κινητοποιήσουμε τις εκθέσεις αυτές και ο μόνος τρόπος να κινητοποιηθούν είναι μέσω του Κοινοβουλίου και γι' αυτό όπως λέω στο σημείο 6 συνιστώ στην Επιτροπή ε, ότι παρόλο που ε, οι η, τροπολογίες υπευλήθηκαν την 1η Δεκεμβρίου ε, ζητείται από την Επιτροπή να αναδιατυπωθούν και να ξαναυποβληθούν τροπολογίες. Η γραμματεία θα μας πει μέχρι πότε θα έχουμε προθεσμία για τις τροπολογίες. Αντιλαμβάνουμε ότι τώρα διακόπτουμε για το καλοκαίρι, αλλά ελπίζω οι τροπολογίες να μπορούν να υποβληθούν σύντομα μετά το καλοκαίρι και στην ε, περίπτωση αυτή θα μπορέσουμε να αντισταθούμε στις πιέσεις του Συμβουλίου διότι νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι συγχωνεύει όλους τους τομείς του θέματος αυτού, ουσιαστικά σε μία πρόταση και αναφέρεται στην περιοχή του Βορείου Βισκαϊκού ε, και είχαμε συζητήσει εχθές ε, την έκθεση αυτή με άλλους συναδέλφους οι οποίοι ανησύχησαν αλλά τους είπα ότι θα επανέλθει το θέμα ενοποιημένο ή στην Επιτροπή μας ότι θα μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε κατά το καλοκαίρι και θα έλεγα να προχωρήσουμε με την έκθεση αυτή να ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο και ελπίζω ότι θα μπορέσει να προχωρήσει στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μπιλμπάου, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος ο φάκελος αυτός από την αρχή. Εγώ πιστεύτηκα την ψήφο προσανατολισμού και όπως ε, εξηγήσαμε στο παρελθόν και στην περίπτωση για το σχέδιο του, απόθεμα, του αποθέματος ε, του Γαύρου, εγώ συνεργάστηκα με τον κλάδο στο Βυσκαϊκό Κόλπο, με τους συνεταιρισμού στη Γαλλικία, μέχρι και ε, του Ιπαράλδε. Οι τροπολογίες που παρουσιάσαμε ανταποκρίνονταν στη συζήτηση και στις πρωτοβουλίες που υλοποιήσαμε με τον τομέα, με τον κλάδο η Επίτροπος Δαμανάκη μας ανακοίνωσε σε μια συνεδρίαση που είχαμε ότι θα παρουσίαζε μια νέα πρόταση που τελικά δεν έφτασε. Και σε μία μετέπειτα συνεδρίαση που υλοποιήσαμε μας ανακοίνωσε ότι δεν επρόκειτο να στείλει μία τροποποιητική πρόταση της αρχικής της Κομισιόν και Παρ' όλα αυτά φαινόταν ε, ότι θα ήταν ανοιχτέ οι πόρτε για να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση με την ψήφο προσανατολισμού που είχε θετήσει η Επιτροπή ελιά. Σε αυτό το διάμεσο χρονικό διάστημα εγώ συναντήθηκα με προσώπους του Συμβουλίου και θεώρησα ότι πάνω κάτω είχαμε μια κατάλληλη συμφωνία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να προβούμε και στον τριμερή διάλογο. Και ενώ προχωρούσαν συζητήσεις με το Συμβουλίο, η Κομισιόν μας έστειλε ένα έγγραφο, ένα, επίσημο έγγραφο, non-paper, το οποίο δεν το καταλάβαμε και πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων μας το έστειλαν. Έτσι λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα εμπόδια, εγώ κάλεσα τον τριμερή διάλογο, και με τις συνεδριάσεις που είχαμε το Συμβούλιο είχα θεωρήσει ότι σε αυτόν τον τριμερή διάλογο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και ότι θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια οριστική ψηφοφορία και να το παρουσιάσουμε στην Κομισιόν. Όμω αυτή την τελευταία συνεδρίαση, όπω είπε και ο Πρόεδρο, το Συμβούλιο μα είπε κατά γράμμα ότι κατόπιν αιτήματο τη κυβέρνηση τη Γαλλία και τη κυβέρνηση τη Ισπανία ε, τελμάτων ο φάκελος γιατί είχαν αμφιβολίες για την νομική βάση. Από τη στιγμή εκείνη μου φαίνεται τρομερό το Συμβούλιο να πρέπει να περιμένει να συγκληθεί ο τρομερής διάλογος να μας ανακοινώσει κάτι τέτοιο. Είμαστε σε παράλυση. Εγώ προσωπικά ε, πιστεύω ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε με τα εργαλεία που έχουμε. Αλλά αναρωτιέμαι χωρίς να έχουμε ακόμη απάντηση από την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου για την κατάσταση. Φαίνεται ότι έχουμε μία έκθεση για το Σαφρίδι και μας δίνουν αρμοδιότητα και αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συναπόφαση. Όμω ε, δεν έχει φτάσει η έκθεση για το Γαύρο, δεν θα έπρεπε να διαφοροποιείται. Αλλά εμένα αυτό που δεν μου αρέσει προσωπικά είναι ε, ότι η Κομισιόν του Συμβούλιο θεωρεί αυτή την έκθεση ουσιαστικό και εγώ θα ήθελα να καλέσω άλλο τριμερή διάλογο για να μπορέσω να προχωρήσω. Αυτό που δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε ως Επιτροπή Αλίας είναι μήπως να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να μας ε, στείλει την έκθεση το συντομότερο και τη συμβιβαστική πρόταση. Γιατί αν δεν έχουμε αυτή τη συμβιβαστική πρόταση, εγώ δεν ξέρω τι δυνατότητε έχουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Η πρόθεσή μου είναι να προχωρήσω όπω το έκανα μέχρι τώρα, αλλά με αυτό το εμπόδιο. Δηλαδή να μην έχουμε ορισμό ή να μην έχουμε γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία και να μην έχουμε και τη θέση του Συμβουλίου. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε ειλικρινά. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάποια προσπάθεια για να ε, ξεκαθαρίσουμε ορισμένα από τα ζητήματα που και η Κομισιόν δεν δέχτηκε και εγκρίθηκαν στην Επιτροπή Αλίας. Εγώ θα ήθελα να προχωρήσω, όμως να μας ξεκαθαρίσει το Συμβούλιο ποια είναι η θέση του, γιατί νομίζω ότι δεν μπορούμε να καθυστερούμε ακόμη περισσότερο τέτοια ζητήματα, τέτοιους φακέλους. A ver, ε, En cualquier caso... Κοιτάξτε, όπω και να έχει σήμερα συζητείτε το θέμα στην Κεροπέρ. Έτσι λοιπόν, ε, δεν γνωρίζουμε ούτε και τι συμβαίνει. Σήμερα συζητείτε το θέμα αυτό, αλλά δεν έχω περαιτέρω πληροφορίε για το περιεχόμενο. Σε πολλούς τομείς Μπορώ να συμφωνήσω με τους δύο εισηγητές, γενικώ όμως θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο ότι θα μπορούσαμε να διορθώσουμε ένα λάθος το οποίο κάναμε κατά την ψηφοφορία σχετικά με την μακροχρόνια διαχείριση του Γαβρού στην τροπολογία 30 αναφερόμασταν σε εγγυημένους 7.000 τόνους ε, και ε, το τονίζω δηλαδή ότι μπορούν να αλλιευτούν 7.000 τόνοι γαβρού πράγμα το οποίο είναι τρέλα κατά τη γνώμη μου. Σας παρακαλώ να με προσέξετε γιατί πιστεύω ότι αυτό μας ε, αφορά όλους. Εάν λοιπόν αποδεχτούμε αυτή την τροπολογία θα μας, ε, ε, θα μας επιπλήξουν διότι πρόκειται για, μια, για ένα τραγικό λάθος και τότε υιοθετήθηκε με μικρή πλειοψηφία στην Επιτροπή. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε το λάθος αυτό και παρακαλώ όλες τις τις ε, πολιτικές ομάδες να συζητήσουν την τροπολογία 30. Το ίδιο αναφέρεται ή ε, στην αύξηση από το 0,3 στο 0,4 δηλαδή ε, ενδέχεται να καταρρεύσει η πιθανότητα αυτή πάρα πολύ εύκολα και επειδή έχουμε κάνει λάθη στο παρελθόν δεν πρέπει να διακινδυνεύουμε Ξέρω ότι οι σοσιαλιστές δεν πρόκειται να υιοθετήσουν την έκθεση αυτή αν δεν διορθωθούν τα θέματα αυτά. Δηλαδή ε, χρειάζεται να διορθώσουμε το πρόγραμμα διαχειρίσεως διότι θα μας επιπλήξουν. Ε, πάντοτε μιλάμε για υπερβολική αλίευση και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Κύριε ρόντου, το θέμα είναι ότι το θέμα αυτό εγκρίθηκε. Το θέμα είναι αν θα ανοίξουμε μια νέα προθεσμία για τροπολογίες. Δεύτερον, πρέπει να σας πω, γιατί εγώ συμμετέχω στις τριμερείς συνομιλίες, ότι το Συμβούλιο ε, συμφωνεί με τις τροπολογίες. Υπάρχει δηλαδή συμφωνία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και η Κομισιόν είναι αυτή που δημιουργεί προβλήματα και εξακολουθεί να διαφωνεί. Ε, δεν ξέρω, μπορεί να έχετε την άποψή σας, αλλά εγώ έχω και τη δική μου άποψη για το πώς έχει το θέμα. κυρία Πατράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ουσιαστικά συμφωνώ με όσα είπαν μόλις οι συζητητές. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα διαδικαστικό πέρα από τα προβλήματα επί του περιεχομένου και θα μπορέσει να αποτελέσει σημαντικό προηγούμενο. Εγώ νομίζω ότι de facto εδώ πρέπει να έχουμε μια κάθετη στάση η οποία να δώσει ένα μήνυμα να προτείνουμε δηλαδή ποια είναι η λύση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πώς θα ασκεί τα καθήκοντά του. Και το να το πράξουμε αυτή τη στιγμή νομίζω είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με έναν τρόπο απόλυτα σαφή σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες ε, του κάθε οργάνου. Έτσι λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πράγματι θα έπρεπε να προχωρήσουμε. Ε, πρέπει να βγούμε από το διέξοδο που έχουμε αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μα ε, και μάλιστα γνωρίζοντα ότι η γνωμοδότηση τη νομική υπηρεσία του ίδιου του Συμβουλίου είναι ουσιαστικά μη ευνοϊκό για το Συμβουλίο και αυτό μα διευκολύνει εμά να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ε, προχωρήσουμε λοιπόν με επίσημη ψηφοφορία, ποιοι είναι στην ίδια των Κομισιόν και να δούμε αν θα πεμπλακεί και σε επίπεδο Συμβουλίου κατάσταση, όπω είπε και ο κ. Γκάλαγκερ, Εμεί θα προχωρούσαμε το Σεπτέμβριο και κατόπιν ε, υπάρχει και αυτή η περίοδος αναμονής που θα επιτρέψει στο Συμβούλιο να λάβει θέση και να δει πώς έχει η κατάσταση κατόπιν της έκδοσης της νομοδότησης της νομικής υπηρεσίας ίσως θα μπορούσε να λάβει μια ευρύτερη θέση συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν το Σεπτέμβριο θα μπορούσαμε να προβούμε στην ψηφοφορία στην Επιτροπή και στη συνέχεια ίσως ε, να ήταν ε, δυνατό με διαφορετική θέση του Συμβουλίου να καταλήξουμε σε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο καταρχήν να αναλάβουμε τις αρμοδιότητές μας ε, και να καθορίσουμε με σαφήνεια ποια είναι η θέση μας ε, και για αυτή την έκθεση, για το Σαφρίδη και για το γάβρο, γιατί είναι ίδια η κατάσταση και φυσικά όλα αυτά θα μας εξυπηρετήσουν και για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν δύο θέματα και νομίζω ότι λίγο πολύ συμφωνούμε για το πρώτο θέμα, ως προς τη διαδικασία δηλαδή. Συμφωνώ με τις προτάσεις που έγιναν, δηλαδή να προχωρήσουμε αναλαμβάνοντας τις δικές μας ευθύνες και κατά κάποιο τρόπο χωρίς να είμαστε αρνητικοί, αλλά να έχουμε μία ε, ανάγνωση από πλευράς Κοινοβουλίου για το πώς ε, ορίζονται τα θέματα αυτά στη συνθήκη της Λισαβόνας. Συμφωνώ με τα αυτά που πρότεινε λοιπόν η κυρία Πατρό Νέβες και οι δύο εισηγητές ε, να προχωρήσουμε και να ακολουθήσουμε τα, αυτά, τις διαδικασίες όπως πρέπει. Όπως είπε ο κύριος Γκάλακερ βέβαια, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία ως πρέπει. Αν πρέπει να κάνουμε και μία ψήφο προσανατολισμού για να δώσουμε μία σαφή εντολή στους δύο εισηγητές, και έγινε λοιπόν και αυτή η ψήφος, αυτή η ψήφος ανατολισμό. Ήδη ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας και πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία όπως πρέπει και νομίζω ότι η πρόταση του κυρίου Γκάλαγκερ είναι σωστή. Να ξεκινήσει η ομαλή διαδικασία, δηλαδή να ξεκινήσει μια προθεσμία τροπολογιών, να παρουσιαστούν οι τροπολογίες, να ψηφίσουμε και αυτό είναι η διαδικασία πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου. Το λέω γιατί θα ήταν περίεργο να κάνουμε όλα αυτά, δηλαδή να ξεκινήσει μια προθεσμία τροπολογιών και για την άλλη να μην το κάνουμε γιατί θα έχουμε ψήφο προσανατολισμό. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν όλα σωστά, δηλαδή από τώρα και στο εξή να ξεκινήσει η προθεσμία για τις τροπολογίες και να προχωρήσουμε όπως προχωράει η Επιτροπή. Για το Σαβρίδι όχι και τόσο, αλλά για το Γάβρο είναι προφανές ότι στο διάστημα αυτό είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση η ψήφος προσανατολισμού που είχαμε τότε για κάποια θέματα, και κάποιος ε, το επεσήμανε εδώ, δεν ήταν ομόφωνη. Δηλαδή έγιναν κάποιες συζητήσεις εις βάθος και θα έπρεπε να ε, συζητήσουμε και κάποια θέματα κλειδί εδώ. Για παράδειγμα, το 30%, το 40% των αποθεμάτων βιομάζας. Ε, ή το όριο του ΤΑΚ ε, αν θα πηγαίνει σε 7.000 τόνους ή θα πρέπει να πάμε κάτω από το 25% όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το 10% που εγκρίθηκε όταν ψήφισε το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει τέλος πάντων όλα αυτά τα θέματα να τεθούν εκ νέου επιτάπητος, να τα ψηφίσουμε και να δούμε ε, τι έγινε και τότε που τα είχαμε συζητήσει στην Επιτροπή. Επιμένω όμως, το πρώτο βήμα είναι να καθορίσουμε μια προθεσμία για τροπολογίε και να ακολουθήσουμε τις ομαλές διαδικασίες ε, των κοινοβουλευτικών εργασιών και ως προς τη συζήτηση, εάν γίνει, κάποιοι από εμά θα θέσουμε κάποια θέματα ουσίας, διότι υπάρχουν ε, κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ομόφωνα από πλευράς Επιτροπής μας. Θα ήθελα να ζητήσω να να δούμε καταρχάς τη διαδικασία και το πώς φτάσαμε ως εδώ. Διότι αν αρχίσουμε να μπλέκουμε τα πράγματα, τελικά στη μία έκθεση μας ενδιαφέρει το ένα και στην άλλη το άλλο. Το βασικό θέμα λοιπόν είναι η διαδικασία. Η κυρία Αντρές Μπαρέα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι ακούω τόση ώρα όλους όσους μίλησαν και νομίζω ότι αυτό το θέμα υπερβαίνει και την ίδια την Επιτροπή. Υπάρχει θέμα αρμοδιοτήτων. Ε, υπήρξε και μια συνεδρίαση με τον κύριο Γκάλαγκερ, είτε είναι για αυτή την έκθεση όμω, είτε είναι για το Γαύρο. Ε, το θέμα που μα ενδιαφέρει είναι η θεσμική αρμοδιότητα που έχει ο καθένα. Ε, φαίνεται να μην τηρεί κάποιο τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ο καθένα θέλει να τηρεί τι εξουσίε του που είχε και πρέπει να το λύσουμε το θέμα αυτό. Κάθε θεσμικό όργανο, δεν ξέρω αν υπάρχει η έκθεση του Κοινοβουλίου, αλλά κάθε θεσμικό όργανο θα κάνει τα καθήκοντά του βάσει της ε, και αυτά θα τα ακολουθεί ο καθένα μέχρι να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητα μόνο τη Επιτροπή Αλία. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο πάει παραπέρα ε, ε, και αν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτά που πρέπει να κάνουν τα τρία θεσμικά όργανα βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα πρέπει να το λύσουμε. Πέραν αυτού όμως, επειδή είναι πολύ δύσκολο να το λύσουμε και είναι πολύ περίπλοκα κάποια πράγματα και ορισμένες φορές ε, οι εκθέσεις ε, καθορίζονται ad hoc ανάλογα με το που ανήκουν, η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι η εξή. Η Επιτροπή μα πρέπει να συνεχίσει τι εργασίε τη και επομένω πρέπει να γίνονται οι εκθέσει βάσει των προθεσμών που καθορίζονται, παρουσιάζονται τροπολογίε και κατά κάποιο τρόπο πιέζοντας με έμεσο τρόπο το Συμβούλιο και την Κομισιόν να προσαρμοστούν και να ε, προχωρήσουν τη διαδικασία. Πέραν του να αποφασίσουμε λοιπόν τα εκ των έσω, δηλαδή το να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και για τις δύο εκθέσεις κατ' Ε, και να καθορίσουμε μια στρατηγική, θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα και σε ανώτερο επίπεδο. Αν εμεί είμαστε η μόνη επιτροπή που έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή με αυτέ τι δύο εκθέσει, τότε έχει Δεν νομίζω όμω να είναι έτσι. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ επιτροπέ που έχουν προβλήματα με την εφαρμογή τη συνθήκη Λισαβόνα. Θα τα πάμε λοιπόν σε ανώτερο επίπεδο για να δούμε τι λύση θα υιοθετήσει το Κοινοβούλιο για την εφαρμογή τη συνθήκη Λισαβόνα. Ωραία. Είναι θέμα της αλληλείας όμως. Είναι θέμα κατανομής αρμαδιοτήτων στον αλληλευτικό τομέα. Ε, τα πάντα είναι συναπόφαση με εξαίρεση τα τάκια της ποσοστώσης και εδώ φυσικά είναι και το πρόβλημα. Εδώ είναι το Συμβούλιο που προσπαθεί να ε, διαγράψει το Κοινοβούλιο, να του πει ότι δεν έχει αρμοδιότητα και προς το παρόν η νομική υπηρεσία μας υποστηρίζει. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα επιλύσουμε, δεν θα χρειάζεται να προσφύγουμε στο δικαστήριο, με την εν ναι, εξαίρεση το Συμβούλιο να εγκρίνει τα πάντα με βάση το 43 το και να μας απορρίψει τελείως. Ε, προτείνω λοιπόν εμείς να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης χωρίς να περιμένουμε συμφωνία με το Συμβούλιο. Εμεί ε, θα προχωρήσουμε, θα παρουσιάσουμε τροπολογίε. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να μπλοκάρει το θέμα ή να μην το μπλοκάρει. Τέλος πάντων, εμείς θα προχωρήσουμε σε πρώτη ανάγνωση χωρίς να έχουμε καταλήξει συμφωνία με το Συμβούλιο ε, και αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία θα πάμε στη δεύτερη, στη ε, συνδιαλλαγή, σε ό,τι χρειαστεί τέλο πάντων. Αποφασίζουμε ότι περνάμε σε διαδικασία πρώτης ανάγνωσης, ό,τι και αν γίνει, ή η άλλη επιλογή είναι να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Κορεπέρ και με το Συμβούλιο αυτές τις μέρες. Ε, αύριο θα έχουμε και εκπρόσωπο της Προεδρίας εδώ, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι και να υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Αυτές είναι οι δύο εναλλακτικέ λύσεις. Αν δεχτούμε την πρώτη, καθορίζουμε ε, ε, προθεσμίες για τροπολογίες. Αν δεχτούμε τη δεύτερη εναλλακτική, περιμένουμε μέχρι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να ξεμπλοκάρουν το θέμα, εκτός και αν το Συμβούλιο πει ότι θα τηρήσει το 43-3, το οποίο και επομένω θα πρέπει και εμεί να προσφύγουμε στο δικαστήριο. Θα δώσω το λόγο στου εισηγητέ και μετά θα λάβουμε απόφαση. Πρώτο είχε ζητήσει το λόγο η κυρία Μπιλπάου και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλαχερ. Να διευκρινίσω το εξή. Όταν είπα ότι πρέπει να προχωρήσουμε, αυτό για μένα σήμαινε δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς ε, την έκθεση της νομική υπηρεσίας του Συμβουλίου και την άποψη του Συμβουλίου για να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε ή όχι. Εάν η άποψη του Συμβουλίου δεν είναι σαφής και κάνουμε άλλη μια άλλη συνεδρίαση και ξεκινήσει μια διαδικασία προθεσμία για τροπολογίε, θα είμαστε στην ίδια κατάσταση. Εγώ προτείνω να διευκρινιστεί η θέση του Συμβουλίου και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε και θα είναι πιο γρήγορη η επίτευξη συμφωνία. Διότι θα έχουμε μια συμφωνία στην οποία θα υπάρχουν διαφορέ που επιτρέπεται να έχουμε. Αυτή είναι η διαδικασία που έχουμε δεκτεί. Το αντίθετο θα ήταν να προκύψει και το ερώτημα γιατί χάσαμε τόσο χρόνο αν τα είχαμε κάνει όλα στο τέλος του χρόνου, τρέχοντας με την ψήφα προσανατολισμό και 1η Ιανουαρίου να είχαμε ξεκινήσει από την αρχή. Ε, ο, αν φτάσαμε μέχρι εδώ ήταν γιατί όλοι είχαμε δεχτεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η διαδικασία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία ίσω θα πρέπει να δεχτούμε για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτό που δεν δέχομαι είναι να παρουσιάζεται ω επιχείρημα το θέμα τη ομοφωνίας. Διότι αν αρχίσουμε να συζητάμε ομοφωνίε και αρχίσουμε να ξαναβλέπουμε τι συμφωνίε κάθε ε, επιτροπή του Κοινοβουλίου αναθέμα, νομίζω ότι τελικώ δεν θα έχει εγκριθεί τίποτα. Εγώ Ω διαδικασία δέχομαι ότι ε, είχαμε πει ότι η ψήφο προσανατολισμού αρκεί και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ζητήσουμε διευκρινήσει από το Συμβούλιο και να διευκρινίσουμε το θέμα για να προχωρήσουμε. Εγώ δεν θα ήθελα να ξεκινήσουν προθεσμίε για κατάθεση τροπολογιών εάν δεν είναι να καταλήξουμε πουθενά. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, να συνοψίσω. Καταλαβαίνω ότι εσεί ω εισηγήτρια θέλετε να συνεχίσετε ω έχει κατάσταση. Δεν θέλετε να πάμε σε πρώτη ανάγνωση πριν να φτάσουμε σε πρώτερη συμφωνία με το Συμβούλιο. Γιατί οι δυνατότητε είναι να φτάσουμε σε πρώτη ανάγνωση είτε με συμφωνία ή χωρί συμφωνία. Εσεί πάντω θέλετε να περιμένουμε να δούμε την γνωμοδότηση τη ε, νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και ανάλογα με αυτό να λάβουμε απόφαση. Συγγνώμη, συνοψίζω, συνοψίζω για να είναι σαφή τα πράγματα για όλους. Κύριε Ρωμέρο, σας παρακαλώ μην με κοιτάτε έτσι. Θέλω απλώς να συνοψίσω τι είπε η κυρία εισηγήτρια, έτσι ώστε όλοι να συμφωνήσουμε και να είναι όλα κατανοητά. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Μπιλμπάου. Sí, ε, Κοιτάξτε, εμεί ε, μπορούμε να πετύσουμε μια στάση από το, Συμβούλιο, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πάρει μια κάποια στάση το Συμβούλιο που θα το πετύσουμε εμεί. Τώρα το θέμα είναι ότι το Συμβούλιο καθυστερεί γιατί θέλει να κερδίσει χρόνο και αυτό χρονοτριβεί. Εγώ τώρα τι να σα πω, μπορώ να πω στο Συμβούλιο ό,τι θέλετε, αλλά τι να σα πω, δεν νομίζω ότι θα κάνουν και κάτι. Κύριος Γκάλακερ. Uh, Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν, όταν συζήτησαμε την, ε, με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρούσαμε γρήγορα, είχαμε φτάσει σχεδόν το ο στόχο μας και τώρα η κατάσταση έχει ατονίσει. Ε, αν ε, ε, δεν είχαμε εμεί όμως αναλάβει την πρωτοβουλία τίποτα δεν θα γινόταν. Τώρα βέβαια κατά τύχη βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξαναλάβουμε την πρωτοβουλία, να ξεκινήσουμε περίοδο τροπολογιών για να κινηθούμε για να μπορέσει, ίσως δεν μπορέσει το Συμβούλιο να καταλήξει σε συνένεση, αλλά εμείς δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τι θα κάνουν οι άλλοι, αλλά τι θέλουμε εμείς και ε, θα πρέπει να ε, σκεφτόμαστε το μέλλον της αλληλείας και αυτής της Επιτροπής. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Ε, και η ε, γνωμοδότηση που έχει λάβει το Συμβούλιο δεν ήταν αυτή την οποία επιθυμούσε. Οπότε δεν μπορεί όλα να τα έχουν. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε και συμφωνώ με την άποψη της Επιτροπής και ε, ό,τι αποφασίσει η Επιτροπή, εγώ απλούστατα θα φροντίσω να το εξυπηρετήσω. Ευχαριστώ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα και δεν μπορούμε να συζητάμε αιωνίως αυτό το θέμα. I agree. Ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Γκάλαχερ ότι πρέπει να καθορίσουμε μία ημερομηνία για τροπολογίες και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Sí, que ya la να σας δώσω σε εσάς το λόγο και στους εισηγητές σας έκαναν λόγο. Η κυρία Πάρο. Ναι, κοιτάξτε, εγώ θέλω να κάνω μια πρόταση βάση και το όσων είπατε εσείς. Εγώ θέλω να προσπαθήσω να καταλήξουμε σε μια λύση. Θα μπορούσαμε ίσως να θέσουμε μια ημερομηνία για το Σεπτέμβριο, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου και από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρξει απάντηση, να ξεκινήσουμε την εξέταση της έκθεσης ε, και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία με τις τροπολογίες και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να είναι μια ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή ας δώσουμε μια ημερομηνία στο Συμβούλιο στα τέλη Σεπτεμβρίου για να αντιδράσει. Είναι μια πρόταση που καταθέτω εδώ. Bueno, pues, eh... Πρόεδρος. Μάλιστα, καλό μου φαίνεται. Στη συνεδρίαση ε, τέλη Αυγούστου θα ξέρουμε τι θα έχει γίνει με την Κορεπέρ και αύριο θα έχουμε και τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Υπουργό Αλίας της Ισπανίας. Ε, νομίζω ότι οι λοιπόν, επόμενες συνεδρίες που έχουμε είναι περί τα τέλη Αυγούστου. Έτσι λοιπόν, βάσει αυτού θα δούμε αν θα απεμπλοκαριστεί η κατάσταση ή όχι και τι θα κάνουμε με τις έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση και τον Αύγουστο θα λάβουμε μία απόφαση. Ευχαριστώ τους εισήγητες. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης που είναι το σημείο 8, έγκριση των τροπολογιών της σύμβασης ε, της ε, ΝΑΦΟ. Εισηγητής είναι ο κύριος Βαλέσα και να του δώσω το λόγο. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Chciałbym pokrótce zaprezentować mój projekt zalecenia w tej sprawie. Ευχαριστώ. Παρουσιάζω το πρώτο σχέδιο. Η σύμβαση είχε συναυθεί το 1978 στην Οτάβα, ίσχυσε από την 1η Ιανουαρίου 1979 και ε, ο στόχος ήταν ε, να αποφύγει την υπερβολική εκμετάλλευση ε, των αποθεμάτων ψαριών και στη συνέχεια άλλαξε το κείμενο αυτό το 2007 και 2008 έγιναν συνεδριάσεις όπου υπήρξαν σημαντικές αλλαγές και ε, όχι μόνο εις τις συμβάσεις αλλά και στα έγγραφα όπου άλλαξε και η ορολογία για τη διαχείριση των ψαριών. Υπάρχει μία σαφής ε, ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτων σημαίας και κράτων λιμένος και ε, ο προϋπολογισμός και οι συνδρομές επίσης έχουν αλλάξει. Υπάρξει δε ε, ε, μία αλλαγή του μηχανισμού επιλύσεως των διαφορών που προβλέπεται και στα πλαίσια αυτά θα πρέπει εμείς να αποδεχθούμε τις αλλαγές. Προτείνω λοιπόν να ε, χορηγήσουμε την ε, συνένεσή μας στο θέμα αυτό. Επιπλέον όμως θα ήθελα να τονίσω δύο θέματα τα οποία είναι προβληματικά και χρειάζονται την προσοχή μας. Αφενός, ότι τα μέρη εις της ε, συμβάσης ε, θα πρέπει να δεχθούν ε, το κείμενο, αλλά στη μία σύμβαση είναι, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο και στην άλλη το γαλλικό. Το έγγραφο της Επιτροπής για την εφαρμογή στην κοινοτική νομοθεσία έχει ημερομηνία Μάρτιος του 2010. Δηλαδή ε, καταρτίζεται επί δύο χρόνια. Τέτοιες ε, καθυστερήσεις είναι απαράδεκτες. Πρέπει να το τονίσουμε και να περιορίσουμε τον χρόνο αυτό, διότι η διετία είναι υπερβολικά μακρύς χρόνος η ταχύτητα με την οποία έγινε ίσως αιτιολογείται από την σωστή διαχείριση αλλά θα πρέπει το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή να μπορέσουν να συνεργαστούν καλύτερα στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, και αυτό το γεγονός αποδεικνύει ότι στην ε, πραγματικότητα υπάρχουν προβλήματα και θα πρέπει να βρούμε τρόπο να τα επιλύσουμε. Το δεύτερο θέμα, το οποίο είναι προφανές, είναι ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ίσχυσε το Δεκέμβριο του 2009 και η ε, κοινοβουλευτική μας επιτροπή απέκτησε νέες δυνατότητες το δε το οποίο συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι το 2007-2008 εμείς δεν εκπροσωπούμεθα σαν κοινοβούλιο, αλλά τώρα θα συμφωνήσουμε, θυμίζοντας όμως την Επιτροπή και στο Συμβούλιο ποιες είναι οι νομικές επιταγές και ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η δικιά μας εξουσία και σας ευχαριστώ. Η κυρία Τροτμάν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ο συγητής μας εξήγησε θαυμάσια και τα υπέρ και τα προβλήματα της εφαρμογής της συνθήκης και της κατανομής και ισορροπίας των αρμοδιοτήτων και των καθυστερήσεων και προθεσμιών. Πρέπει να σας πω ότι συμφωνούμε με αυτή τη σύμφωνη γνώμη διότι πιστεύουμε ότι οι βελτιώσεις αυτές και ο εξυγχρονισμός της συμφωνίας είναι απαραίτητα θέματα. Πρέπει να αυξήσουμε την αξιοπιστή ε, μας, να επιλύουμε πιο γρήγορα τις διαφορές και η Επιτροπή μας θα πρέπει να τονίσει, όπως είπε ο εισηγητής, τη θέλησή μας να μην υπάρξουν επιπρόσθετες καθυστερήσεις. Εμείς δεν επιβραδύνουμε. Αντιθέτως είμαστε υπέρ μίας επιτάχυνσης των δραστηριοτήτων και συμφωνώ και με την ενέργεια. Το Κοινοβούλιο δηλαδή να συνομιλεί με ένα Συμβούλιο το οποίο θα σέβεται τις αρμοδιότητές μας σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και θα πρέπει να υποφεληθούμε τις ευκαιρίες που μας δίνεται να ε, τονίσουμε το σημείο αυτό σε σχέση με το παρελθόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και κύριε Βαλέσα. Πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως με την ε, γνώμη σας όσον αφορά τις ε, ε, καθυστερήσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες, χρειαζόμαστε να επιταχύνουμε. Έχω όμως μία ερώτηση σχετικά με το περιεχόμενο της νέας συμφωνίας, σχετικά με τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων η οποία αναθεωρήθηκε. Όσον αφορά ε, τις υποχρεώσεις των συμβαλωμένων ε, μερών που θέλουν να εφαρμόσουν μία διάταξη της σύμβασης, δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε, διότι ε, δεν ξέρω εάν μπορείτε κιόλας να το σχολιάσετε. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε, λέει η πρόεδρος, ο κύριος Καντέκ πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, πρέπει να κάνω μια παρατήρηση που συμφωνεί με τα προηγούμενα. Δηλαδή πρέπει να πούμε στον συνάδελφο Βαλέσα ότι έχει δίκιο όταν λέει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για τις επόμενες συμβάσεις γιατί είναι νέες αρμοδιότητες. Βλέπετε ότι σε όλες τις εκθέσεις υπενθυμίζουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας η οποία δεν γίνεται πάντοτε κατανοητή ε, και δεν εφαρμόζεται από όλους. Επίσης έχει δίκιο όταν λέει ότι πρέπει να βελτιωθεί η ε, διαδικασία νομοθετικά για να κερδίσουμε χρόνο και να στηρίξουμε τον συνάδελφο Βαλέσα στις ενέργειές τους και στον τρόπο με τον οποίο να αντεπεξέρχεται του συναχιού από το οποίο πάσχει. Ευχαριστώ κύριε Βαλέσα. Κυρία Πατράου. Eu serei muito breve, eh, apenas para... Πολύ σύντομα. Για να συγχαρώ τον συνάδελφο για το έργο του καταρχήν και να τονίσουμε εδώ μία από τις πτυχές που ήδη αναφέρθηκαν ε, από τους προλαλήσαντες. Δηλαδή την αναγκαιότητα να μην ε, έχουμε καμία καθυστέρηση περαιτέρω της διαδικασίας και ούτε να δεχτούμε τις καθυστερήσεις που θα μας επιβληθούν και επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω την αναγκαιότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι παρόν και να εκπροσωπείται στις διαπραγματεύσεις, να παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις αυτές. Για μια ακόμη φορά, εδώ μιλάμε για νέες διαδικασίες και πρέπει να είμαστε από την αρχή κάθετοι στη στάση μας. Αν εδώ υιοθετήσουμε μία σταθερή, μία κάθετη θέση καθώς έχουμε νέες διαδικασίες βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας. Και αν το πράξουμε αυτό από την αρχή, σίγουρα στο μέλλον θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για μας. Και το ότι είμαστε παρόντες στις διαπραγματεύσεις θα μας δώσει ε, τη δυνατότητα όχι μόνο να έχουμε μια πιο ταχεία διαδικασία, αλλά θα συμβάλλει και στο να έχουμε την οικοδόμηση ευρύτερων συμβιβασμών. Και αυτό είναι ο στόχος όλων των ευρωπαϊκών οργάνων. Έτσι λοιπόν αυτό ήθελα να πω, να έχουμε μια κάθετη στάση στις νέες διαδικασίες συνεργασίας με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα, γιατί αυτό θα αποτελέσει και το μοντέλο για το μέλλον. Ευχαριστώ. Να δώσω καταρχήν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν σε εσά, κυρία Βαλέσα. Ας ακούσουμε καταρχήν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εδώ την εκπρόσωπη της Κομισιόν. Um, thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Κομισιόν θα ήθελα να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την ε, έκθεση αυτή. Όπω είπαμε και στο παρελθόν, η Κομισιόν πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για να, ε, να επικυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι ε, τροπολογίε στη σύμβαση αυτή. Όπω είπατε, πρόκειται και σε ξεχρονισμό του μέσου αυτού και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το υλοποιήσουμε. Να κάνω όμω ορισμένα σχόλια. Τόνισε ο εισηγητής ότι αυτή η διαδικασία δεν ήταν ιδιαίτερα ταχεία. Η Κομισιόν ε, το αναγνωρίζει. Ή, όπως εξήγησε η Κομισιόν κατά την παρουσίαση αυτού του σημείου, είχαμε κάποια νομικά ζητήματα που ανέκυψαν. Η τρέχουσα σύμβαση συνήθει από την Ευρωπαϊκή ανεκυψαν η τρεχουσα συμβαση συνηθι απο την ευρωπαικη κοινοτητα τότε υπό τη μορφή του κανονισμού Συμβουλίου. Ενώ τώρα μιλάμε για απόφαση του Συμβουλίου. Έτσι λοιπόν είχαμε ένα νομικό ζήτημα για το ποιο είναι το σωστό μέσο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και αυτό προκάλεσε κάποιες καθυστερήσεις. Η Κομισιόν δεν είναι ικανοποιημένη φυσικά με κάτι τέτοιο, αν τώρα σας παρηγορώ. Μόνο δύο μέρη αυτή τη σύμβαση ε, έχουν κυρώσει μέχρι σήμερα αυτή τη σύμβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι το τρίτο μέρο που θα το πράξει και θα θέλουμε να σα διασφαλίσουμε. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τέτοιε καθυστερήσει ε, δεν θα λάβουν χώρα στο μέλλον. Η Κομισιόν λοιπόν δεν θεωρεί ότι είναι συστημικό το πρόβλημα, απλώ έτυχε λόγω περιστάσεων. Επίσης, ε, γνωρίζουμε ποιε είναι οι νέε αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη θέση της της Λισαβόνας και φυσικά πρόκειται να σεβαστούμε στο μέλλον τις αρμοδιότητες αυτές κατά γράμμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συμμετείχαν σήμερα στη συζήτηση και να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή σαν Επιτροπή Αλίας μπορούμε είτε να πούμε ναι είτε όχι. Δεν μπορούμε να επισέλθουμε στις λεπτομέρειες και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε περισσότερα να σχολιάσουμε. Ευχαριστώ. Les recuerdo Να σας υπενθυμίσω ότι ήδη επανειλημμένο μέσω της γραμματείας ε, έχει νοσοποιηθεί τροπολογίες για αυτές τις εκθέσεις που βασίζονται σε μια γνωμοδότηση δεν μπορούν να είναι τροπολογίες που να φύγουν ούτε τη συμφωνία του πρωτόκολλο, ούτε τη σύμβαση αλλά πρέπει να αφορούν αποκλειστικά Το είναι νομοθετική απόφαση, νομοθετικό ψήφισμα και όπως ε, ξέρετε η Προεδρία της Κομισιόν κατόπιν ε, ε, φυσικά διαβουλεύσεων με τις νομικές υπηρεσίες θα τις υλοποιήσει τις τροπολογίες αυτές. Τώρα με την αλλαγή με τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες τροπολογίες όπως στο παρελθόν και πρέπει οι τροπολογίες να αφορούν μόνο το ψήφισμα. Δεν μπορούμε να τροπήσουμε τη σύμβαση, ούτε τα πρωτόκολλα, τίποτα. Έτσι λοιπόν, ορίσω τώρα το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση αυτή. 2 Σεπτεμβρίου, προθεσμία για τις τροπολογίες, κατάσταση τροπολογιών, 2 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, 21 Σεπτεμβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή και τον Οκτώβριο θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια, 2 Οκτωβρίου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαλέσσα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και το σημείο 8. Ας περάσουμε στο σημείο 9 της ημερησίας διάταξης που είναι η συμφωνία με τις νήσους Σολομόντος. Η κυρία Πατραονέβες έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρόκειται για μια συμφωνία ελευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των νήσων του Σολομόντος. Είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια συμφωνία έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι για διαβούλευση, όχι δηλαδή για συμβουλευτική τοποθέτηση από εμάς, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε. Και μπορούμε αν και δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε τροπολογίες, μπορούμε όμως να παρουσιάσουμε κάποιες συστάσεις. Κάτι που έγινε στην περίπτωση αυτή. Η συμφωνία αυτή αναφέρεται σε μια αντικατάσταση της προηγούμενης συμφωνίας, η οποία έχει να κάνει με την ελήψη των οειδών και αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση προηγούμενη συμφωνία ίσχυε μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2009 και αυτή η συμφωνία αντικατάστασης ήδη εφαρμόζεται προσωρινά από τις 9 Οκτωβρίου του 2009. Τώρα, οι τροποποιήσεις και να ευστήσω την προσοχή σας εδώ και να σας αναφέρω ποιες είναι οι πιο σημαντικές πτυχές. Μιλάμε για μια χρηματοοικονομική συνεισφορά, η οποία διατηρείται για μια αυξημένη υποστήριξη της ε, τομεακής πολιτικής ε, αλληλείας των νησών της Ολομόντας από το 30% περνάμε στο 50% και η μεγάλη διαφορά θα είναι ότι δεν προβλέπεται πλέον δυνατότητα λίας ε, από τα παραγαδιάρικα επιφανείας. Ε, στο παρελθόν ούτως ή άλλως δεν είχαν χρησιμοποιήσει τις ελευτικές τους άδειε. Αυτό επίσης έχει ως αποτέλεσμα ε, στην αλλαγή των τόνων αναφοράς από τους 6.000 τόνους το χρόνο, περνάμε στους 4.000 τόνους το χρόνο. Και Αυτά προκάλεσαν κάποιες ανησυχίες σε μένα. Τα έχω σημειώσει στην έκθεση που παρουσιάζω. Γιατί έχουμε την ε, ίδια χρηματοοικονομική στήριξη στις νήσους του Σολομόντος ε, σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία, ενώ τώρα μιλάμε για μείωση των ε, αδειών, των ελευτικών αδειών και μείωση και του όγκου των ελευμάτων που επιτρέπεται να ληφθούν. Επίσης, πρέπει να προσθέσω ότι η προηγούμενη συμφωνία από οικονομική σκοπιά δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική. Η αποδοτικότητά της ε, ουσιαστικά βασιζόταν και σε άλλες ε, συμφωνίες για την αλία των, ε, των οειδών. Και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι αυξάνεται αρκετά η συνεισφορά για τους εφαπλιστές. Περνάμε στο 1500 ευρώ τώρα. Η Κομισιόν μας είχε ενημερώσει ότι πρόκειται για έτοιμα των ίδιων των εφοπλιστών αυτό. Τώρα τέλος. Το ότι η Μικτή Επιτροπή Παρακολούθησης δεν έχει συνεδριάσει όπως είχε προβλεφθεί και αυτό είναι ενισχυτικό γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για να χαρακτούν οι άξονες της συνεργασίας. Έτσι λοιπόν τονίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά στο μέλλον. πτυχέ αυτές παρουσιάζονται ω λοιπόν που πρέπει να ληφθούν στο μέλλον και στο παρόν και στο μέλλον. Θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία πάντως πρέπει να υλοποιηθεί για διάφορες πτυχές που επίσης αναφέρονται στην γνωμοδότηση, στην έκθεση. Καταρχήν, αναγκαιότητα να διερευνήσουμε τη συνεργασία σε μια περιφερειακή βάση προκειμένου να πετύχουμε τη βιωσιμότητα πέραν των υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό κρίνεται στη σύσταση τη πράσινη Βίβλου για τη μεταρρύθμιση τη κοινής πολιτική και σε ένα ψήφισμα που υιοθετήθηκε στι 25 Φεβρουαρίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέρα από το να απελθέσουμε ότι η Συμφωνία προβλέπει την πρόθεση της συνεργασία σε αυτή την πλευρά του Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού. Και φυσικά αυτό είναι μία από τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια άλλη πτυχή που πρέπει να αναφέρουμε εδώ είναι ότι η μελέτη αξιολόγησης της συμφωνίας μας έδειξε ότι η διατήρηση των σχέσεων του αλληλευτικού ε, τομέα ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως ε, σε ό,τι αφορά στον εφοδιασμό της δικής μας βιομηχανίας και της κοινοτικής αγοράς. Καθώς ε, εμείς, όπως γνωρίζετε, εισάγουμε πολύ τόνο. Και κάτι άλλο θετικό είναι το ότι οι νήσοι του Σολομόντος ε, χρειάζονται αποθέματα για την μακροοικονομική σταθερότητά τους και αυτή η συμφωνία προβλέπει ότι για τρία χρόνια θα ισχύει και θα δίνεται χρηματοδότηση και αυτή η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της ε, εθνικής τομέκης πολιτικής αλίας. Και αυτό αποτελεί μία από τις αποστολές που αναλαμβάνει τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιοχές αλίας στο εξωτερικό σε αυτή τη συμφωνία αντικατάσταση ε, έχει σαχθεί όχι μόνο μια ρήτρα αναθεώρηση η οποία προβλέπει να υπάρξουν σημαντικοί προσανατολισμοί αλλά υπάρχει και μια ρήτρα διασφάλισης η οποία επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει ε, αν το επιθυμεί, να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να αναστείλει την ε, εφαρμογή του πρωτοκόλλου και να αναθεωρήσει την χρηματοοικονομική συνεισφορά αν αιτιολογείται κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν έχουμε μια συμφωνία η οποία ε, δεν ε, είναι αυστηρή για τα τρία έτη, δηλαδή μας επιτρέπει να έχουμε μια ευελιξία και επιτρέπει μια προσαρμογή κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ετών. Αν ενδεχομένως αλλάξουν οι συνθήκες. Έτσι λοιπόν, η πρόταση που παρουσιάζω εδώ είναι να εγκρίνουμε τη συμφωνία αυτή. Και στο σημείο 2 έχω συμπεριλάβει κάποιες συστάσεις. οι οποίε φυσικά συνάδουν με τα όσα μόλις σας παρουσίασα. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Πατρόν Νέβεθ για την ε, καλή δουλειά που έκανε. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι ανησυχώ για το γεγονός ότι η παλιά συμφωνία η προσωρινή συμφωνία ε, δεν ε, λαμβάνει υπόψη ότι ε, έπρεπε να μην προχωρούμε αυθόρμητα, αλλά πρώτα να διασφαλίσουμε ότι ε, ε, έχουμε καλύψει ε, τα σημεία της συμφωνίας και αυτό το κατακρίνω. Πέραν αυτού όμως, πρέπει να είμαι και λιγάκι κοινικό σχετικά με τις οικονομικές πτυχές, διότι μιλάμε για 1,5 εκατομμύρια ευρώ για 3 εκατομμύρια για τέσσερα πλοία. Δηλαδή ε, θα πληρώσουμε 1,5 εκατομμύριο για τέσσερα πλοία για να λιεύουν επί τρία χρόνια στη νησιά του Σολομώντας. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορώ να το εξηγήσω στους ψηφοφόρους. Στο παρελθόν ήταν 14 τα πλοία Οπότε ήταν διαφορετική κατάσταση. Είμαι και στην Επιτροπή Προπολογισμού. Έχει γίνει μία δήλωση την οποία διαβάσατε και είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι αυτή η συμφωνία είναι καλή. Δεν είναι καλή συμφωνία. Έχω σπουδάσει ε, οικονομικά και πρέπει να σας πω ότι αυτή δεν είναι καλή επιχείρηση, είναι μια πολύ κακή επιχείρηση. Ε, και ε, ίσως διαβάζετε ε, τα σχόλια της Επιτροπής Ανάπτυξης σχετικά με αυτό το θέμα το οποίο είναι πολύ, κατακρίνει πολύ την κατάσταση οπότε δεν μπορώ να αντιληφθώ πόσο θα εφαρμόσουμε τις συστάσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης διότι δεν ξέρω αν η επόμενη συμφωνία θα μπορέσει να ε, υλοποιηθεί. Οπότε, παρόλο που συμφωνώ με την σωστή προσέγγιση του εισηγητή, πρέπει να σας πω ότι κατακρίνω πάρα πολύ. Επίσης, όσον αφορά όλες αυτές τις αλλιευτικές συμφωνίες, οι οποίες καταρτίστηκαν μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας μπορούν τώρα να κατακριθούν και από πλευράς οικονομικής και ε, λόγω του ότι η συμφωνία αυτή όντως δεν αποδίδει όπως θα έπρεπε, δεν προσφέρει ε, οικονομικά ωφέλη ε, και στις δύο πλευρές ή τουλάχιστον μπορεί να προσφέρει στους άλλους και όχι σε εμά. Ε, και δεν νομίζω ότι έχουμε ενημερωθεί επαρκώς για τις λεπτομέρειες. Σαν εισηγητής δεν νομίζω ότι προχωράμε και πιστεύω ότι κανείς άλλος εδώ δεν ξέρει ακριβώς πού κατευθυνόμαστε. Διαφωνώ με τον κύριο Χάγκλαντ. Νομίζω ότι η οικονομική προσέγγιση είναι πολύ σωστή ο κύριος Αρσένης, διότι πληρώνουμε 400.000 το χρόνο, τουλάχιστον για 4.000 τόνους αλλιεύματα και ε, σημαίνει ότι πληρώνουμε 100, το, 100 ευρώ τον τόνο ενώ η τιμή είναι αστρονομικά υψηλότερη οπότε για, ε, για εμάς αυτά είναι πολύ λίγα χρήματα και ε, στηρίζουμε έναν αλλιευτικό στόλο εδώ είναι μια επιλογή την οποία έχουμε κάνει και οι ε, ε, ε, αλείς πληρώνονται 13 ευρώ τον τόνο και αλλάζει το ποσό εάν ξεπεράσουν τις 4.000 τόνους. Ε, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι ουσιαστικά είναι απεικιοκρατία, δηλαδή δεν τους πληρώνουμε τίποτα για αυτό το οποίο μας αποδίδουν και αυτό μας ενδιαφέρει και μας επηρεάζει όλους. συζητάμε μία τώρα συζητάμε μία έκθεση η οποία είναι μία συμφωνία που ισχύει ήδη από τις 9 Οκτωβρίου 2009 και πιστεύω ότι ακόμη και αν είναι μεταβατική περίοδος δεν μπορεί να συνεχίσει, δηλαδή ε, δεν μπορεί το κοινοβούλιο να είναι αφανές στο μέλλον, δεν μπορούμε να ε, συζητάμε αυτές τις συμφωνίες εάν ε, δεν έχουμε έναν ουσιαστικό ρόλο. Δεν είμαστε διακοσμητικά πρόσωπα, ε, συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων. Οπότε είναι κάτι που συζητήσαμε και στην Επιτροπή Ανάπτυξης διότι ε, το γεγονός είναι ότι η Κοινή Επιτροπή ποτέ ε, δεν συνεδρίασε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσωπήθηκε εις την Επιτροπή Ανάπτυξης όταν το συζητήσαμε και μας είπε ότι το έχουν συζητήσει και θα, το, θα θέσουν το θέμα. Πιστεύουμε ότι καλύτερα ε, να, ε, να ψαρεύει στην περιοχή αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι κάποιος άλλος. Ε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει βάση ορισμένων αρχών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει κυρία Ανδρέας Παρέα. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τη συμφωνία που έχουμε. Συμφωνώ απολύτως με την εισηγήτρια, με τα όσα μας είπε και με τις συστάσεις της. Θα ήθελα εδώ όμως να επισημάνω το εξής. Αυτό δεν αποδίδει εισοδήματα και δεν αποδίδει εισοδήματα διότι ο στόχος είναι η ανάπτυξη των νησιών του Σολομόντος και όχι μόνο η ανάπτυξή τους αλλά και ο στρατηγικός ρόλος που έχει ο ε, Ανατολικός Ειρηνικός και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται συνολικά στην αλία τον κόσμο και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη διατήρηση και την εκμετάλλευση των ε, ειδών. Δεν έχω πληροφορίες για την προηγούμενη συμφωνία, αλλά βάσει και της, ε, αυτής της συμφωνίας θα έχουμε και επιστημονικά κριτήρια και όχι μόνο για τον ερυθρό τόνο, αλλά και για άλλα είδη που έχουν σημασία. Υπάρχει κοινωνικός ρόλος στην περιοχή για την ανάπτυξή της και κυρίως, κυρίως υπάρχει ενδιαφέρον διότι ο χώρος ο οποίος καταλαμβάνουμε εμείς με τα κριτήρια της βιωσιμότητας, ε, κριτήρια της ε, διατήρησης των αλευμάτων, κριτήρια της ανάπτυξης της περιοχής, ε, θα είναι ένας χώρος στον οποίο δεν θα μπορούν να έλθουν άλλοι αλληλείς, ε, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ιαπωνία που είχαν τα νησιά του Σολομόντος ως φέουδο. Εάν δεν υπογράψουμε εμείς τη συμφωνία με τα νησιά του Σολομόντος, θα έρθουν οι ΙΠΑ και η Ιαπωνία και θα ε, κάνουν εκμετάλλευση με άλλα κριτήρια τα οποία δεν θα λαμβάνουν σίγουρα υπόψη τους στο περιβάλλον αλλά και άλλους παράγοντες. Σε πολλές από αυτές τις συμφωνίε, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με κυβερνήσει που είναι πολύ περίπλοκες και που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και είναι πολύ δύσκολο να τηρήσουν ε, και τις ε, ρήτρε που περιλαμβάνουν οι ίδιε οι συμφωνίε. Χαίρομαι ε, που υπάρχει μια ρήτρα διασφάλισης εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και η ρήτρα αναθεώρηση επίση, και θα πρέπει εδώ να φροντίσουμε να τηρούνται οι συμφωνίες και να λογοδοτούν για όλα και Θεωρώ ότι είναι γεωστρατηγική σημασία στο να είμαστε παρόντες ε, στον Ανατολικό Ειρηνικό για την ίδια την περιοχή, για την ανάπτυξή τη, με βάση και τις κοινωνικές τη συνθήκες, αλλά και για να σεβαστούμε τα περιβαλλοντικά στοιχεία. Πρόκειται για μια συμφωνία που θεωρώ ότι πρέπει να υπογράψουμε και θα πρέπει να την ενδυναμώσουμε. Ναι, μεν είναι 400.000 ευρώ, αλλά αυτά τα, αυτό το ποσό είναι σημαντικό για την περιοχή, γίνεται μια αλλαγή και από 30% που είχαμε στην προηγούμενη συμφωνία, το 50% πλέον των κολληδίλειων διατίθεται για την ανάπτυξη τη περιοχή και αυτό καταδεικνύει κάτι και είναι πάρα πολύ σημαντικό να την υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία λοιπόν. Η κυρία Λεβίν. Thank you very much and thank you, Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Διάβασα τη, τα συμπεράσματα και την αξιολόγηση για τις σχέσεις μεταξύ ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, νήσων του Σολομώντα και αναφέρεται στο σημείο 13 ότι η συμφωνία απέτυχε διότι παρόλο στους όρους συμφωνίας και του πρωτοκόλου. Η Κοινή Επιτροπή δεν μπόρεσε ποτέ να συναντηθεί από τις εφαρμογές του πρωτοκόλου και δεν μπόρεσε ποτέ να καθορίσει τα συστατικά της συνεργασίας για να υπάρξει μία προώθηση των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ενότητας. Και αυτό υποδηλεί ότι συνδρομή ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 120.000 ευρώ ετησίως έχει χρησιμοποιηθεί για άλλους στόχους. Δηλαδή, προφανώς αυτή η συμφωνία συνεργασίας δεν έχει ακόμη αποδώσει. Και με τα χαράς βλέπω ότι υπάρχει κάποια βελτίωση με τη νέα συμφωνία όσον αφορά την ε, ρήτρα αναθεώρησης, αλλά τίποτα δεν με ε, πείθει ότι η ανάπτυξη και το τμήμα της συρρήξεως του τομέα λαμβάνεται στα σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι θα εξασφαλιστεί ότι τώρα θα εφαρμοστεί ότι οι κοινέ επιτροπές συνεδριάζουν, διότι ούτε οι τεχνικές επιτροπές δεν έχουν συνεδριάσει στα τρία χρόνια από τη σύναψη συμφωνίας. Όταν βλέπω και τα αποθέματα που αναφέρονται στην αξιολόγηση, υπάρχει αναφορά τον, στα αποθέματα του, του τόνου, ενώ δεν ε, πρόκειται ε, για καθαρό τόνο, πρόκειται ε, ε, για ε, λακέρδα ή για άλλα είδη τόνου και έχουμε στοιχεία ότι θα πρέπει να υπάρξει μείωση της αλίας διότι υπάρχει υπερβολική. Επίσης ένα άλλο πράγμα το οποίο με ανησυχεί είναι ότι δεν υπάρχει ένα πλαφό και υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής αδειίας ε, στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ για να διατηρηθεί η συμφωνία και σύμφωνα με την αξιολόγηση είναι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να υπάρχει ένα πλαίσιο πολιτικό ώστε να υπάρξει μία βελτίωση. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω πιστεί από αυτά που άκουσα ότι η νέα συμφωνία θα αξιοποιήσει τα σωστά στοιχεία. Και προσωπικά είμαι πολύ επιφυλακτική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στίβενσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αναμφισβήτητα χρειαζόμαστε τα ψάρια στην Ευρώπη, είναι προφανές και συμφωνώ με τον κύριο Αρσένη ότι δεν είναι και κακή οικονομική συμφωνία. Συμφωνώ επίσης με τον κύριο, ε, την κυρία Άντες Βαρέα ότι εάν εμείς αποσυρθούμε άλλοι θα εκμεταλλευτούν τα, ε, τα ψάρια αυτά και ε, δεν θα σκεφτούν καθόλου πώς θα διατηρηθούν τα αποθέματα λίας. Πρόσφατα όμως είχαμε πάει στην επιθεώρηση αλία στο Βίγκο και μας ελέγχθη ότι υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς αυτές τις συμφωνίες τις αλλιευτικές εάν υπάρξει επαρκής ε, χρηματοδότηση. Έχουμε δει την αποτυχία των ε, προηγουμένων συμφωνιών με τις Νιούς Σολομόντα όπως είπε η προλαλήσασα. Ξέρουμε ότι σε πολλά θέματα υπήρξε υπεραλίευση ή τα χρήματα δεν χρησιμοποιήθηκαν για την ε, συντήρηση των αλλιευτικών πόρων και σήμερα το απόγευμα που θα μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό θα πρέπει να ε, συζητήσουμε τον κύριο Κώστα και να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά μας όταν γίνονται τέτοιες ε, συμφωνίες διότι χρειαζόμαστε ε, τους πόρους διότι υπάρχει οικονομική κρίση εάν όμως θέλουμε να διατηρήσουμε τα διεθνή αλληλευτικά αποθέματα είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Επίσης ε, ε, έχουμε έναν ενισχυμένο ρόλο στη σχέση με αυτές τις συμφωνίες χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας και πριν από χρόνια ε, είχαμε ζητήσει ένα μέλος της Επιτροπής να συμμετέχει σε όλες τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη αυτών των ε, συμφωνιών και μας είχαν κλείσει την πόρτα ε, στα μούτρα. Τώρα όμως δεν μπορούν να το κάνουν, οπότε καλό θα ήταν ένα μέλος αυτής της Επιτροπής να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις όλων αυτών των συμφωνιών κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε επισέλθουμε αυτών των δυσκολιών τις οποίες αντιμετωπίζουμε και δεδομένων των σωστών απόψεων της Επιτροπής θα πρέπει να επέμβουμε στις διαπραγματεύσεις για να προχωρήσει σωστά το όλο θέμα. Ευχαριστώ. Όλα αυτά είναι πολύ σωστά. Δεν θέλω εδώ να αναφερθώ στο περιεχόμενο των συμφωνιών, απλούστατα να διευκρινίσω ότι εδώ σύμφωνα με τις τελευταίες διαβουλεύσεις δεν θα έχουμε δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε μία μικρή, μεικτή επιτροπή γιατί αυτό έχει απορριφθεί. Το ξέρουμε από την Επιτροπή Συντονιστών και ίσως εδώ θα έπρεπε να μας πει ο υπεύθυνο τι έγινε στις διαπραγματεύσεις, διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε. Και νομίζω ότι υπήρξαν πολλές φάσεις όπου θα έπρεπε να έχουμε συζητήσει αν μπορούμε να δεχθούμε αυτή την αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι και στο μέλλον δεν πρόκειται να ε, παριστάμεθα στις διαπραγματεύσεις ε, που θα διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, έπρεπε σαφώς να πούμε ότι ε, η συνθήκη της ε, Λισαβόνας δεν ε, εφαρμόζεται σωστά. Θα έπρεπε να συμμετέχουμε και να τους πούμε ότι δεν θα συνενούμε σε αυτές τις αλλιευτικές συμφωνίες αν δεν έχουμε συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Να αποφασίσουμε λοιπόν σήμερα ότι δεν θα αποφασίσουμε επί του θέματος σήμερα αλλά θα ξανασυζητήσουμε και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να εκπροσωπήσω εν ανάγκη όλη την πολιτική μου ομάδα αλλά δεν μ' αρέσει να με σπρώχνουν έτσι νομίζω ότι δεν πρέπει να το δεχτούμε γιατί θα μας περιμένουν μαύρες μέρες συνέχεια Κύριε σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα σύντομο σχόλιο στους φίλους μου Κρήτων και Στέρεν για το κατά πόσον είναι καλή συμφωνία. Σαφώς είναι καλή συμφωνία για την Αλία, αλλά είναι χειριστικά και στη συμφωνία για τους φορολογούμενους. Ε, αν ήμουν εγώ ένα από αυτού που είχε τα τέσσερα λιευτικά σκάφη, θα ήμουν εξαιρετικά ικανοποιημένο. Αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση καλή συμφωνία για τους φορολογούμενους, φίλοι μου. Εγώ θα ήθελα να πω ένα-δύο πράγματα, λέει ο πρόεδρο. Τα θεσμικά νομίζω ότι τα συζητήσατε όλοι και θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε κάλλιστα και σε άλλη στιγμή. Καταρχά, θα ήθελα να πω ότι αυτή η περιοχή του Ειρηνικού που μα ανησυχεί ω προ του πόρου τη, είναι αντικείμενο διαχείριση μια περιφερειακή οργάνωση αρία, ε, η Επιτροπή ε, του Δυτικού και Ανατολικού Ειρηνικού. Δεν δίνονται περισσότερε άδειε από αυτέ που δίνονται μέσω αυτή τη περιφερειακή οργάνωση ε, του ε, δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού ε, και υπάρχουν κάποια θέματα που επισήμαναν κάποια, τα είδαμε και στην έκθεση της Μικτής Επιτροπής, το θέμα της ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη. Και είναι αλήθεια, υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να επιλύσουμε. Και είναι αλήθεια ότι είναι και εξαιρετικέ οι συνθήκε, αλλά είναι εξαιρετική και η τοποθεσία στην οποία βρίσκονται τα νησιά του Σουλομόντου. Πρόκειται για μια χώρα η οποία είναι σε διαδικασία ανάπτυξη. Να σα δώσουμε ένα παράδειγμα μια χώρα που βρίσκεται πιο, ε, είναι κοντά και έχουμε συμφωνία με αυτήν, το Κυριμπάτι. Και εδώ θα πρέπει να σα υπενθυμίσω ότι ε, εγώ ήμουν αρμόδια για την υπόθεση. Χρειάστηκε να περιμένουμε από το Μάιο, διότι το Κυριμπάτι έχει τόσο πολλά νησάκια και για να συναντηθούν χρειάζεται να συναντηθούν επισήμω μία φορά το χρόνο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα νησιά του Σολομόντος, αλλά με τον Κυριμπάτι τα ξέρω τα πράγματα και υπάρχουν και τέτοιες δυσκολίες. Έχει δίκιο ο κύριος Στίβενσον όταν λέει ότι όταν συζητάμε τον προπολογισμό, ένα από τα θέματα στα οποία έγιναν ε, πολύ μεγάλες περικοπές ε, το Συμβούλιο είναι αυτές οι γραμμές προπολογισμού που γίνονται για να ε, καταβληθούν τα έξοδα ταξιδίου αυτών των φτωχών χωρών που δεν έχουν χρήματα για να έρθουν στις μεικτές επιτροπές. Και αυτό φυσικά το ξεχνάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έγινε τεράστια περικοπή σε αυτά τα κονδύλια. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τώρα για τι συμφωνίε αλλήλίε ότι πρόκειται για κοινή πολιτική. Τα ίδια πράγματα έχουμε με την Γεωργία, αλλά ε, η διαφορά είναι ότι πολύ θα ήθελα εγώ να έχω τα χρήματα που έχει η Γεωργία. Είναι κοινή πολιτική αλληλεία ε, σχόλιο εκτό μικροφώνου του κ. Χάγκλοντ, δηλαδή θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν έχουμε κοινή πολιτική, η χρηματοδότηση κυρίω προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα αρέσει, δεν μα αρέσει, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Τώρα, ω προ τη χρηματοδότηση, θα ήθελα να πω απλώ το εξή λησμονούμε ότι από αυτό το κεφάλαιο υπάρχει ένα τεράστιο τμήμα το οποίο δίνεται για την ανάπτυξη και υπάρχει και ένα σημαντικό τμήμα το οποίο ε, είναι ε, για τους ε, κοινοτικούς πλειοκτήτες. Και υπάρχει κάτι το οποίο δεν ανέφερε κανεί από του παρόντε και αυτή είναι η έκθεση αξιολόγηση και θα ήθελα να θέσω την ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση αξιολόγηση συστήνει όλε αυτέ τι συμφωνίε του κεντρικού, αρενικού και όλη τη περιοχή, το Κυριμπάτι και όλε τι υπόλοιπε περιοχέ, έχουν μείνει ουσιαστικά στα χέρια του Θεού γιατί είναι πάρα πολύ μακρινέ. θα έπρεπε ίσω να υπάρχουν κάποιοι αρμόδιοι που θα ασχολούνται με αυτά τα θέματα του ειρηνικού, να δει τι δυσκολίε υπάρχουν και να ασχοληθεί με τα θέματα τη εξέλιξη και τη ε, υλοποίηση αυτών των συμφωνών. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο θα λάβει υπόψη τη ε, η Επιτροπή αυτή την παρατήρηση που έχουμε στην έκθεση αξιολόγηση. Έχουμε και άλλε συζητήσει οι οποίε μπορεί να είναι ίσονο σημασία, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω εάν η Κομισιόν ε, έχει σκοπό να κάνει κάτι, διότι πράγματι αυτέ οι χώρε βρίσκονται πάρα πολύ μακριά και είναι αφημένε στο έλεο του Θεού. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω εάν σκοπεύετε να κάνετε κάτι. Ο κύριος Κάτεκ θέλει το λόγο. Όχι, δεν πρόκειται να μιλήσω μετά από εσά. Δεν ήθιστε, Πρόεδρε. Απλώ ε, ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την εισηγήτρια και ότι πρέπει να εγκρίνουμε την συμφωνία με τις νήσους του Λεμόντος, αλλά οι συνάδελφοι ουσιαστικά τοποθετήθηκαν και είπαν τα ουσιαστικά πράγματα που έπρεπε να αποθούν. Ευχαριστώ, κύριε Αλεξάνδρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να επανέλθω σε ορισμένες αντιδράσεις πολύ ενδιαφέρουσες οι οποίες αναπτύχθηκαν από τους αξιότιμους ευρωβουλευτές. Δεν ε, θέλω να επενέσω το νέο πρωτόκολλο, αλλά ορισμένες από τις παρατηρήσεις οι οποίες διατυπώθηκαν ε, πρέπει να λάβουν απάντηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχήν, Ορισμένοι από εσά ε, ίσως εκπλήσονται ότι με μία μείωση του, της τονοχωρητικότητας αναφοράς και μείωση των αδειών αλληλείας ε, για τα πλοία έχουμε τον ίδιο οικονομικό φάκελο ο οποίος όμως διαμορφώνεται διαφορετικά διότι έχουμε μετατοπίσει περισσότερη χρηματοδότηση εις ε, την ε, πολιτική, τομεακή πολιτική της αλληλείας. Και αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερον, νομίζω ότι η κυρία Πατράο Νέβες στην ομιλία της μίλησε για τη σημαντική αύξηση ε, της ε, συνδρομής ε, των πλειοκτητών στο πρόγραμμα παρατηρητών. περάσαμε από 400 σε 1500 ευρώ. Ήταν μια σύσταση η οποία διατυπώθηκε από την ε, ε, η ε, εντόπια επιτροπή ε, αλληλεία στην περιοχή για τον τόνο που προβλέπει να υπάρχει ε, κάλυψη 100% των εξόδων και προσπαθήσαμε να διατυπώσουμε μία σύσταση κατόπιν ε, αυτής ε, της αποφάσεως του τοπικού οργανισμού. Όντως αυτό το ζήτησαν οι νήσοι του Σολομόντος και ε, συμφωνήσαμε Έπρεπε λοιπόν η διμερή συμφωνία μας να αντικατοπτρίζει αυτήν την σύσταση. διότι δεν είχαμε καμιά αντίρρηση ουσιαστικά. Πολλοί ευρωβουλευτές πολύ σωστά ανέφεραν και ε, επαναλαμβάνω αυτό που είπα πέρυσι στην Επιτροπή Ανάπτυξης ότι κατά τα τρία τελευταία έτη η μεικτή ε, επιτροπή που προβλέπεται εις το πρωτόκολλο δεν έχει συνέλθει. Ε, δεν είπα ότι σοκαριστικά ο κύριος Αρσένης χρησιμοποίησε τους ίδιους όρους με μένα, αλλά είμαι υπεύθυνο ε, για την μονάδα αυτή από την 1η Δεκεμβρίου και είπα ε, σε όλους τους συνεργάτες μας ότι πρέπει να σεβαστούμε όλες τις υποχρεώσεις που αναγράφονται στα πρωτόκολλα και ένα από αυτά είναι να υπάρξουν κοινέ μικτές επιτροπές και αν χρειαστεί θα πάμε στο τέρμα του κόσμου ώστε αυτή η ετήσια υποχρέωση να συνέρχεται η μικτή επιτροπή να μπορέσει να εφαρμοστεί. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο από κοινού θα αξιολογήσουμε ε, την ε, συγκεκριμένη υλοποίηση και την χρησιμοποίηση συγκεκριμένα από την τρίτη χώρα επί του προκειμένου της νήσου του Σολομώντα των ποσών που τους διετέθησαν ε, στα πλαίσια της συμβάσεως και για να γίνει μια κοινή αξιολόγηση των αλλιευμάτων και του σεβασμού από τους πλειοκτήτες των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει. Ε, δεν θα ήθελα λοιπόν επουδενή λόγο οι συμφωνίες αυτές ε, να αποτελέσουν ε, αντικείμενο μη σεβασμού διότι έχουμε ε, ε, ε, έχουν όλοι οι στόλοι ατέλειες αλλά εμείς προσπαθούμε να ελέγχουμε καλά και θα θέλαμε οι υποχρεώσεις να γίνονται σεβατές από όλους συμπεριλαμβανομένων και των πλειοκτητών των αλλιευτικών. Δεν θα επανέλθω στα θεσμικά θέματα τα οποία έθιξαν συνάδελφοι. Ξέρετε τώρα υπάρχει η συνθήκη της Λισαβόνας και υπάρχει διαφορετική ρύθμιση των συμφωνιών μας. Είμαστε δε έτοιμοι να ακολουθήσουμε το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα ήθελα όμως να επανέλθω εις ε, το, την πτυχή των οικονομικών που ανέφεραν διάφοροι. Δηλαδή ότι πληρώνουμε για τέσσερα πλοία και ουσιαστικά τους δίνουμε 400.000 ευρώ ετησίως. Επανέρχομαι όμως αυτά που είπα πέρυσι στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα τέλος πρόσβασης, δικαίωμα πρόσβασης. Γι' αυτό πληρώνουμε, για να έχουν τέσσερα κοινοτικά πλοία δικαίωμα πρόσβαση διότι δεν αλλιεύουν ευτυχώς μόνο εις την ε, ζώνη των ε, νήσων του Σολομόντος αλλά και στον Ειρηνικό, στην ανοιχτή θάλασσα και ε, σε άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες. Αυτό ήταν όμως πολύ βασικό να τονιστεί διότι δεν πληρώνουμε ε, τα αλλιεύματα, πληρώνουμε απλούστατα ένα δικαίωμα πρόσβασης και υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι δυνατότητες ε, αλλιευμάτων δεν ε, χρησιμοποιούνται διότι οι πλειοκτήτες δεν θέλουν να πάνε εκεί. Και αυτό είναι διαφορετική συζήτηση. Κυρία Πρόεδρε, εσείς αναφερθήκατε σε μία από τις δυσκολίες της υπάρξεως αυτών των συμβάσεων που βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου σε σχέση με την Ευρώπη και προτείνατε να υπάρξει μία ενίσχυση προσωπικού στις αντιπροσωπείες μας που θα μπορούσε να παρακολουθεί εκ του την ε, εξέλιξη αυτών των ε, συμφωνιών, να συμμετέχει στις τεχνικές συζητήσεις και να συμμετέχει με τους εκπροσώπους των ε, Βρυξελών στις μικτές επιτροπές. Το ξέρουμε, το προβλέπουμε, διότι αν θέλουμε να διατηρήσουμε την παρουσία μας, ιδίως στον Ειρηνικό ωκεανό, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις επιτόπου αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που μας απασχολεί και ελπίζουμε ότι αρκετά σύντομα θα τελεσφορήσει. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ όλους τους ευρωβουλευτές που έλαβαν το λόγο και είμαι στη διάθεσή σας για να σας απαντήσω. Ευχαριστούμε κύριε Αλεξάνδρου. Λοιπόν, να ορίσουμε την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. 2 Σεπτεμβρίου. Συγγνώμη, η συγγήτρια, η κυρία Πατράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, όντω ήθελα το λόγο. Να ξεκινήσω καταρχήν ευχαριστώντα τον εκπροσωπό τη Κομισιόν για την παρεμβασή τη, ε, για τι πτυχέ που εκφράστηκαν εδώ Όλα όσα είπατε είχαν ε, ήδη υποθεί κατά την παρουσίαση της έκθεσης ε, και το ότι από 400 ευρώ περνάμε στα 1500 και αυτό ήταν έτοιμα ε, των ίσων. Παρουσιάζονται λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα μάλα, τις παρατηρήσεις, τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Και να σας πω ότι κατά κάποιο τρόπο ήδη συμπεριλαμβάνονταν ε, στην έκθεση που παρουσίασα. Αυτό σημαίνει ότι το ισοσύγιο, δηλαδή η αποτίμηση που έκανα και τελικά ε, το ότι συστήνω την έγκριση της συμφωνίας αυτής ε, σημαίνει ότι δεν αγνοούμε τις θετικές πτυχές. Και εδώ Στη σύσταση έχω συμπεριλάβει και ένα σημείο 2. Δηλαδή να υιοθετηθεί μία θέση κάθετη και να ζητήσουμε μία νέα διαδικασία από την Κομισιόν. Έτσι λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτό το θεσμικό ζήτημα είναι θεμελιώδες. Και το ξαναλέω. Όταν ε, συζητήσαμε τη γνωμοδότηση Βαλέσα, εγώ τόνισα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα είναι παρόν και θα παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις. Για μια ακόμη φορά και πάλι αιτιολογείται εδώ κάτι τέτοιο. Εγώ θεωρώ και επαναλαμβάνομαι τώρα ότι υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να εγκρίνονται, να υιοθετούνται ταχαίως, με σταθερό τρόπο, έτσι ώστε αποφεύγουμε προβλήματα να αποφεύγουμε προβλήματα στο μέλλον. Μπορούμε να είμαστε παρόντες και να παρακολουθούμε τη διαδικασία. Το ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι αυτό και το είχα πει και εγώ. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το περιεχόμενο. Αυτό καθ' αυτό. Να σας πω ότι φυσικά και εγώ συνορίζομαι πολλές από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν εδώ, αλλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήδη είχαν συμπεριληφθεί στο κείμενο που σας παρουσίασα. Η αλήθεια είναι ότι, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις τυχές εδώ, πρέπει να δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζει μια θεμελιώδη θέση σε αυτή την περιοχή, γεωστρατηγική θέση. Έχει σημασία να τη διατηρήσουμε. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι αν εμείς δεν υπογράψουμε τη συμφωνία να αποσυρθούμε θα παραμείνει κενός ο χώρος αυτός. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με τους όρους αυτούς όπως υπόθηκε, άλλοι θα έρθουν με άλλα κριτήρια, πολύ χειρότερα από τα δικά μας, που δεν θα έχουν τις δικές μας βαλίστες πρακτικές και δεν έχουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το χώρο. Έτσι λοιπόν, Όντω, συμμερίζομαι ορισμένε από τι ανησυχίε που ακούστηκαν εδώ. Ακούσαμε και τη συζήτηση για το αν είναι καλή ή κακή η συμφωνία. Όμω πρέπει να το δούμε όλο αυτό το θέμα συνολικά. Και εγώ θεωρώ, και αυτή είναι η θέση μου, γιατί θεωρώ ότι αυτή η πτυχή υπερισχύ των υπολείπων πρέπει να διασφαλίσουμε τη θέση μας σε αυτή την περιοχή. Γιατί πρόκειται για στρατηγική περιοχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ε, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των ίσων του Σολομόντος, γιατί εμείς έχουμε πολύ πιο αυστηρά κριτήρια από οποιοδήποτε άλλη χώρα του κόσμου και Επομένως, θα πρέπει να διατηρηθεί η θέση αυτή. Θα πρέπει να την υπερασπίσουμε αυτή τη θέση εμείς. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι με όλες τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν εδώ και με ακούσαμε από την ε, Επιτροπή, θα πρέπει για την μελλοντική ε, εκπόνηση νέων συμφωνιών, θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει αυτά να τα έχουμε κατά νου, αλλά δεν θα πρέπει να διακινδυνεύσουμε αυτήν εδώ τη συμφωνία, η οποία είναι θεμελιώδης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θεμελιώδης και για τις νήσους του Σολομόντος και πρέπει να λάβουμε εδώ μια υπεύθυνη θέση, να μην αγνοούμε κάποιες πτυχές οι οποίε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για μελλοντική αναθεώρηση όχι μόνο αυτή τη συμφωνία, αλλά όλων των συμφωνιών. Και αναφέρουμε συγκεκριμένα στην αναγκαιότητα του να συνεδριάζει η Μεκτή επιτροπή για να παρακολουθεί όλη αυτή τη διαδικασία και να έχουμε και εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλε αυτέ τι διαδικασίε. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι προκύπτουν πάρα πολύ σημαντικά θέματα από αυτή τη συζήτηση και ξεπερνούν ούτω ή άλλω το περιορισμένο χώρο αυτή τη συμφωνία. Εγώ νομίζω λοιπόν, αν δούμε συνολικά το ζήτημα, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε αυτή τη ε, συμφωνία, γιατί θα είχαμε σε αντίθετη περίπτωση πολλά μειονεκτήματα και ζημιέ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τι ίδιε τι νήσου τη Ολομόντα. Κοιτάξτε, έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Η κυρία Ρουμπούστα έχει ζητήσει το λόγο. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επαναληφθώ εδώ. Κυρία Πατραονέβες, θα έχετε δίκιο. Όντω θα έπρεπε να συμμετέχουμε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να εμπλακούμε γιατί αυτές οι αποφάσεις έχουν δηληφθεί. Αναμένω να μας πει η κυρία Φράγκα πώς θα εργαστούμε στο μέλλον, αλλά εγώ έχω την ε, εντύπωση ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε σε αυτές τις μικτές επιτροπές. Πρέπει να στείλουμε τώρα ένα μήνυμα, γιατί κανένας δεν θα μας πάρει σοβαρά διαφορετικά. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να το πράξουμε, κυρία Φράγκα. Όπως είπα και στους συντονιστές, ε, θα μιλήσω για αυτό το θέμα, όμως ε, τώρα έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Αύριο θα αναφερθώ σε αυτό το θέμα, αλλά τώρα πρέπει να συνεχίσουμε με την ημερησία διάταξη, γιατί διαφορετικά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Κυρία Πατράο. Λοιπόν, 2 Σεπτεμβρίου για τις τροπολογίες, 29 Σεπτεμβρίου για την ψηφορία στην Επιτροπή. Κυρία Ρουμπούστ. Äh, Κυρία Φράγα, με συγχωρείτε, αλλά αύριο δεν έχουμε συνεδρίες των συντονιστών, άρα δεν θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και είχα ζητήσει να καταρτήσουμε μία ομάδα εργασίας η οποία θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό, δηλαδή τι θα κάνουμε στο μέλλον με τις ε, ε, συμφωνίες ε, αλίας, διότι δεν συμμετείχαμε στο παρελθόν και θα παρακαλούσα να ψηφιστεί η πρότασή μου. περίεργος Κοιτάξτε, εγώ είπα ότι θα κάνω την πρόταση και θα την υποβάλω ψηφοφορία. Το θέμα είναι ότι όμως τώρα δεν προλαβαίνουμε. Θέλω να συνεχίσω με την ημερησία διάταξη. Εγώ σας υποσχόμαι ότι αυτό το θέμα θα το δούμε και θα του αφιερώσουμε το χρόνο που το αξίζει, όχι σε αυτό όμως το σημείο γιατί ε, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις συμφωνίες ε, και με τις διαδικασίες μας. υπόσχομαι ότι αύριο θα το ξαναδούμε πλήρως το θέμα αυτό. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στο σημείο 10 της ημερησίας διάταξης, κανόνες για την εισαγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λευτικών προϊόντων, ζώντων θεωρομαλακίων, εχινόδερμων, κοιτονόζων και θαλάσσιων καστερόποδων. Λοιπόν, για τι ε, τροπολογίες 2 Σεπτεμβρίου, ψηφοφορία 29 Σεπτεμβρίου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια Οκτώβριο 2. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στο σημείο 10 της σημερινής διάταξης. Ε, δεν θα επαναλάβω τώρα τον τίτλο. Λοιπόν, με την Γρυλανδία, όπως γνωρίζετε, εδώ συμπεριλαμβάνονται ο κατάλογος ε, των χωρών. Έχουμε το παράρτημα 2 της συνθήκης και σύμφωνα με το άρθρο 198 της συνθήκης, ε, ο στόχος είναι η προώθηση των, ε, της ανάπτυξης των υπερπόντιων χωρών, των υπερπόντιων εδαφών. Εδώ λοιπόν συνάπτουμε μια συμφωνία μεταξύ Γρυλανδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπάρξει μια υγειονομική συμφωνία για τα ζώτα δίθυρα μαλάκια, χινόδερμα, χιτονόζια, θαλάσσια γαστερόποδα αλλά και τα υποπροϊόντα τους. Ο στόχος είναι η Γρυλανδία να μπορεί να ανταλλάσσει αυτά τα προϊόντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και αυτό είναι το σημαντικό. Φυσικά, πάντοτε αφού η Γρυλανδία σεβαστεί την υγειονομική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό η ε, αρχή υγειονομική και διατροφική ε, αρχή της ε, Δανίας και η αρμόδια αρχή της Γρυλανδίας θα είναι αρμόδιες αρχές και θα είναι υπεύθυνε για την εφαρμογή της συμφωνίας. Εγώ πρέπει να σας πω ότι εδώ είπε κάτι η Κομισιόν που με ανησύχησε την τελευταία φορά ότι εξακολουθούμε να είμαστε πολύ μακριά από το η να σεβαστεί όλη την νομοθεσία και είπαν με ακρίβεια ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα πριν η κοινότικη νομοθεσία να μπορέσει να εφαρμοστεί πλήρως από την πλευρά της Γρυλανδίας. Και Τέλος, έχουμε και μία μικρή λεπτομέρεια που είναι το πρόβλημα της νομικής βάσης. Εμείς ε, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει ε, ισχύσει το άρθρο 43 της συνθήκης καθώς στο πρωτόκολλο της Γρυλανδίας λέγεται ότι όλα αυτά τα μέτρα σε σχέση με τις εισαγωγές προϊόντων θα έπρεπε να εφαρμοστούν βάσει του άρθρου 43 και δεν έγινε κάτι τέτοιο ενώ ε, αυτό το άρθρο της συνθήκης που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 203. Έτσι λοιπόν, εγώ θέλω να σε επισημάνω ότι γνωρίζουμε ότι για το θέμα αυτό δεν έχει γίνει σεβαστή η νομική βάση, όμως καθώς είχαμε πάρα πολλά προβλήματα με τις νομικές βάσεις, όπως έχουμε με όλα τα πολιετή σχέδια, αποφασίσαμε και το αποφασίσαμε και στους συντονιστές, να μην κάνουμε τίποτα με το θέμα αυτό, γιατί ε, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στο 10 ε, κατά τη συμβουλή κτλ. Έτσι λοιπόν απλώς είπαμε ότι δεν συμφωνούμε με τη νομική βάση και θεωρούμε ότι κάποια στιγμή αυτό το θέμα θα πρέπει να βασίζονται στο άρθρο 43. Θα πρέπει να έχουν αυτό ως νομική βάση. Τώρα, από την πλευρά της Κομισιόν της ΓΔ ΣΑΝΚΟ έχουμε εδώ την κυρία Στρίκλαν. Εκεί είναι. Les doy δώσω το λόγο. Tiene usted la palabra. Thank you very much, Adam. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όπως πολύ σωστά επισημάνατε, πρόκειται για μια συμφωνία μάλλον μία απόφαση που βρίσκεται στο πεδίο εφαρμογής της ε, Γρυλανδίας, θεωρείται ένα από τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπατε και εσείς οι ίδιοι έχουμε υποχρέωση να αναπτυχθούν οι περιοχές αυτές και να έχουμε στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ ε, ημών και των περιοχών αυτών. Επίσης υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου από το 2006 που δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, βοηθήσει στην ανάπτυξη της Γροιλανδία και να ε, προάγει κυρίως τα θέματα της διατροφικής ασφάλειας. Και αυτό ακριβώς κάνει αυτή η συμφωνία. Επιτρέπει στη Γρυλανδία να τοποθετήσει αλληλευτικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά βάσει των κανόνων ε, τους οποίους υποχρεούνται να τηρήσουν τα κράτη-μέλη, επομένως συμμετέχει στην εσωτερική αγορά δεν υπάρχει καμία ε, επιπλοκή από οικονομικής πλευράς, δεν υπάρχουν δασμοί ε, ή αλλαγές σε ποσοστά οι οποίες θα προκύψουν από αυτή την απόφαση. Η προτινόμενη απόφαση σχετίζεται απλώς ε, σε μέτρα υγεία, με μέτρα υγείας, αλλά θα διευκολύνει τα κάποια θέματα, διότι δεν θα υπάρχουν ανάγκη για πιστοποιητικά εξαγωγών, δεν θα πρέπει να υπάρχουν κατάλογοι από πλευράς επιτροπής και ούτω καθεξής επειδή αναφερθήκατε στην νομική βάση, θα ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι που ακούω ότι θα συζητήσετε το θέμα αυτό σε άλλη περίπτωση, διότι εγώ δεν είμαι αρμόδια για να επισέλθω στα θέματα της νομικής βάσεως, αλλά σαφώς θα μεταβιβάσω το μήνυμα ότι σας ενδιαφέρει το θέμα αυτό και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ όσων βλέπω δεν υπάρχουν και πολλές ερωτήσεις, επομένως θεωρούμε ότι ε, έλεξε το θέμα, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών ε, στις 7 ε, Σεπτεμβρίου, ψηφοφορία 29 Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια θα περάσει τον Οκτώβριο. Σας ευχαριστώ. Ήσασταν νομίζω και στο γραφείο του κυρίου Μπόργκ, οπότε σας γνωρίζουμε μέσω του γραφείου του κυρίου Μπόργκ. Συγχαρητήρια λοιπόν για την νέα σας θέση και σας εύχομαι και καλή τύχη στην Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Και με αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι έληξε το σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης και περνάμε στο σημείο 11, ενδιάμεση συμφωνία εταιρική σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ε, του Ειρηνικού και η συγγήτρια είναι υποφαινόμενη όχι γιατί είναι πρόεδρος της Επιτροπής αλλά γιατί αυτό αποφάσισε η πολιτική μου ομάδα. Ο, η επί Επιτροπή είναι η Επιτροπή Ίντα και εμείς απλώς θα συντάξουμε μια γνωμοδότηση. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η συμφωνία ήδη εφαρμόζεται προσωρινώς από τον Ιανουάριο φέτος και ο στόχος της συμφωνίας είναι να επιτρέπεται η πρόσβαση στην κοινοτική αγορά με πολύ ε, ευνοϊκές προϋποθέσεις ε, κάποιων προϊόντων, αλληλευτικών ε, και κατά βάση μας ενδιαφέρει ο τόνος εδώ, αναφερόμαστε στον ειρηνικό και μας ενδιαφέρουν δύο χώρες κυρίως, η Παππούα Νέα και τα και Τα η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης με πρώην χώρες ΑΚΕ, ε, μόλις έχουν καθορίσει τις εμπορικές συμφωνίες βάσει της Συμφωνίας της Κοτονού. Και γι' αυτό ακριβώς αυτές οι πρώην ΑΚΕ ε, υπογράφουν συμφωνίες ε, οικονομικής σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αντικατάσταση των συμφωνιών που είχαν υπογράψει μέσω της Συμφωνίας του Κοτονού. Θα ήθελα απλώς για να μην ε, πω πάρα πολλά πράγματα, να πω ποιο είναι το βασικό πρόβλημα από πλευρά αλληλεία που διαπιστώνουμε σε αυτή τη συμφωνία. Και το πρόβλημα είναι ότι για πρώτη φορά, ή μάλλον σχεδόν για πρώτη φορά, υπάρχει πλήρης παρέκκληση από μία, για μία από τις ε, ιερές ε, συμφωνίες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα υπάρχουν παρεκκλήσει για πολύ απλά ε, προϊόντα, όπως για παράδειγμα παράγωγα τόνου, και θα υπάρξουν πολύ αρνητικέ συνέπειες και για την ε, κοινοτική βιομηχανία του τόνου, αλλά και για χώρες ε, ΑΚΕ, οι οποίες μέσω κοινοτικών επενδύσεων με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν πάρα πολλές ε, Επενδύσει. Για την Παππούα Γουινέα και τα νησιά Φίτζη δεν έχουμε καμία θέση. Πρόκειται για ανταγωνιστέ μα ουσιαστικά. Οι Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες είναι αυτέ οι οποίε θέλουν να διαδραστηριοποιηθούν στην Παππούα Νέα Γουινέα. Διότι η Παππούα Νέα Γουινέα δεν έχει στόλο και γι' αυτό θεωρείται ότι ε, παρακάμπτονται οι κανόνες ε, προέλευσης. Ποιες είναι οι κανόνες προέλευσης για να μην υπάρχει πρόβλημα. Μία πρώτη ύλη έχει προέλευση, για παράδειγμα, από την Παππούα Νέα Γουινέα ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν, για την περίπτωση της αλίας, αλλιεύεται από σκάφη της παππού Νέας Γουινέας σε ε, ύδατα της οικονομικής ε, αποκλειστικής ζώνης ή σε διεθνή ύδατα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θεωρούμε ότι έχουμε τόνο για παράδειγμα προέλευσης παππού Νέα Γουινέας. Για τα μεταποιημένα προϊόντα που θα διευκρινίσουμε αργότερα ότι είναι τα προϊόντα που μας ενδιαφέρουν κυρίως σε αυτή τη συμφωνία μιλάμε για προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ε, πρώτες ύλες προέλευσης από την παππού Νέα με, σε ένα ποσοστό που επιτρέπει ένα 15% ε, μέγιστο να προέρχεται από άλλη χώρα. Για παράδειγμα, κονσέρβα τόνου θεωρούμε ότι είναι προέλευση της Νέας Γουινέας όταν ε, το 85% είναι τόνος από την Παππούα Νέα Γουινέα. Η παρέκκληση τώρα προκύπτει διότι η Παππούα Νέα Γουινέα δεν έχει στόλο. Και ε, στην έκθεση αποτίμηση αντικτύπου που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία διάβασα αναλυτικά και θα την επικρίνω αργότερα, λέγεται ότι επειδή τα νησιά Φίτζη και η Παππούα Νέα δεν έχουν στόλο, ε, ισχύει παρέκκληση για τους κανόνες προέλευσης. Ποιος όμως επωφελείται από την παρέκκληση αυτή για τους κανόνες προέλευσης και τι συνέπειες μπορεί να έχουν η παρέκκληση σαφώς ε, αφορά τους δικούς μας ανταγωνιστές, οι οποίοι βρίσκονται επιτόπου στην περιοχή και μιλάμε και πάλι για τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη και μόλις έμαθαν ότι θα συμβεί αυτό, άρχισαν μαζική ανάπτυξη ε, σε όλη για παράδειγμα την ακτή του Αντούν που είναι εκεί που γίνεται η ε, παραδοσιακή αλληλεία και ε, χρησιμοποιούν τον όρο Pacific Marine Industrial Zone. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα δούμε αργότερα και τι επιπτώσεις υπάρχουν από κοινωνικής πλευράς. Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω, για να καταλάβετε καλά πώς λειτουργεί όλη η διαδικασία, ότι ο κατεψυγμένος τόνος ως πρώτη ύλη έχει ε, κατόφλι 0 και υπάρχουν κατόφλια για εισαγωγές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κονσέρβες τόνου. Σε αυτή την περίπτωση, με αυτή τη συμφωνία, δίνεται 0% κατόφλι και για τις κονσέρβες τόνου που είναι προέλευσης ε, Παππούας Νέας Γουινέας, δηλαδή ουσιαστικά στους ανταγωνιστές μας, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη. Την ξεχνάω συνέχεια την Ταϊλάνδη, αλλά ε, τέλος πάντων ουσιαστικά τους δίνουμε τη δυνατότητα να εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με δασμό 0. Πρόκειται για συμφωνίες που είχαμε με ε, χώρες ε, πρώην ε, ΑΚΕ, στις οποίες έγιναν επενδύσεις για να τους βοηθήσουμε στον τομέα αυτό. Ακούγεται ένα πουλί, τι είναι αυτό και λαϊδάει κάτι η έκθεση για τα θέματα της, ε, του τόνου ε, στο Κυριμπάτι, στην Παππούα Νέα και λοιπά χώρες δηλαδή που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας λέει ότι οι κοινωνικές επιπτώσεις των επιχειρήσεων τόνο δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη. Οι μισθοί που καταβάλλονται στους εργαζόμενους είναι κατώτεροι από τους απαραίτητους για να μπορέσουν να συντηρήσουν την οικογένειά τους και ε, δεν βοηθά φυσικά τους εργαζομένους να διαφύγουν της ένδυας. Ε, επιπλέον αυτές οι βιομηχανίες και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται και με τις δικές μας ε, μεταποιητικές βιομηχανίες ε, ε, και με τις βιομηχανίες στην Ταϊλάνδη που εισάγουν, διότι το εισάγουν, το λέω εδώ, διότι βρίσκονται σε συνθήκες ε, δουλείας, δουλείας τους πληρώνουν 60 ευρώ και ε, τους δίνουν απλώς τροφή και στέγη. Το ίδιο ακριβώ γίνεται και στην Παππούα Νέα Γουινέα. Ουσιαστικά λοιπόν οι κοινωνικές επιπτώσεις και η βοήθεια στην ανάπτυξη αυτών των πληθυσμών είναι το, αν μη τι άλλο ελληματικέ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνεται τίποτα για αυτέ τι χώρε, αλλά το θέμα είναι ότι οι περιβαλλοντικέ κοινωνικέ και οικονομικέ επιπτώσει για την ανάπτυξη τη παππού νέα Γουινέα είναι πολύ περιορισμένε. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα αρνητικό γιατί κάποιο θα το εκμεταλλευτεί. Θα ήθελα επίση να πω ότι πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσεις και έχω πάρα πολλέ πληροφορίε από του γιατί με ενδιαφέρει πέραν των περιβαλλοντικών προβλημάτων για την ανάπτυξη της ε, ακτής ε, στην οποία γίνεται κυρίως η αλίευση ε, και η εκμετάλλευση εργατικού δυναμικού σε πολύ επισφαλείς συνθήκες όπως σας είπα, υπάρχουν και θέματα παιδικής εργασίας. Και σας το λέω εδώ, όχι γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη χώρα στην οποία υπάρχει, υπάρχουν παιδιά που εργάζονται, αλλά γιατί όντως ισχύει. Και τέλος υπάρχει και ένα ε, σημαντικό πρόβλημα και στο αναφέρω τελευταίο και μας ενδιαφέρουν όλους ε, τα θέματα παράνομης και λαθρέας αλληλείας και εδώ έχουμε παράνομη και λαθρέα αλληλεία. Μιλάμε για μια περιοχή του Ειρηνικού που όπως είπαμε πριν και στα νησιά του Σολομώντα υπάρχει συγκεκριμένη κατανομή των ε, επιτρεπόμενων αλλευμάτων ε, διότι υπάρχει περιφερειακή οργάνωση που διαχειρίζεται τα ίδια αυτά και καθορίζει ποια θα δίνονται. Και θα ήθελα εδώ να σας πω για παράδειγμα ότι δημιουργούνται και νέε νέες εγκαταστάσεις, ε, τρία νέα από, την, από τις Φιλιππίνες, μία από την Ταϊλάνδη και μία νέα από την Κίνα και θα ήθελα να ξέρω τι πόρους θα εκμεταλλευτούν. Δεν είναι πολύ δύσκολο να ε, πούμε ότι υπάρχει ανησυχία, ότι μπορεί να υπάρχει παράνομη λαθρέα και άναρχη αλληλεία, διότι εδώ υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, όλες οι αλευτικές δυνατότητες έχουν κατανεμηθεί, επομένως τι πρώτη θα χρησιμοποιήσουν αυτές οι νέες εγκαταστάσεις. Ποιος θα μας το πει εδώ ότι το, το θέτω ως ερώτηση γιατί δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ λογικό συμπέρασμα. Α, και να μην ξεχάσω, η προβλεπόμενη παραγωγή, για να έχετε και αυτό το στοιχείο, για τα επόμενα δύο χρόνια είναι 426.000 τόνους κονσέρβα που είναι ουσιαστικά το διπλάσιο αυτού που παράγει ε, ένας από τους μεγάλους παραγωγούς, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, σε δύο χρόνια υπολογίζεται να έχουμε αυτό το στοιχείο, το οποίο πήρα από τις πληροφορίες που μου έδωσαν, αυτό υπολογίζεται ότι θα παραχθεί στην περιοχή. Να σας πω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ήρθε εδώ να μας ενημερώσει αναφέρθηκε σε μια διάσημη περιβόητη μελέτη αντικτύπου. Γνωρίζετε πολύ καλά πώς γίνονται αυτές οι μελέτες αντικτύπου. Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου είπε ότι έκανε δική της μελέτη αντικτύπου για τα θέματα αλίας. Εγώ διάβασα λοιπόν αυτή τη μελέτη αντικτύπου η οποία λέει ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αντίστοιχο κλάδο. Βέβαια, κάποιο πρέπει να μα το αποδείξει αυτό. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν επαληθεύουν όλε τι πληροφορίε που έχω εγώ από άλλε πλευρέ. Αυτή η μελέτη αντικτύπου μου φαίνεται απλώς βασική, δεν εμβαθύνει σε τίποτα και δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτά όλα τα οποία δηλώνεται στη μελέτη σα. Επιπλέον, στη συμφωνία εκεί που μιλάμε για τις ε, παρεκκλήσεις για τις χώρες ε, προέλευσης, προβλέπεται και μία αναθεώρηση σε τρία χρόνια. Δεν θα πω εγώ εδώ ότι δεν πρέπει να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, γιατί όλα αυτά είναι έτοιμα. Ε, το επισημένο όμως αυτό, και το επισημένο διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά για τι πράγμα σας μιλάω, θα ήθελα να ζητήσω, εάν συμφωνείτε, από την, Ευρωπαϊκή, από, συγγνώμη, από την Επιτροπή ΙΝΤΑ, πριν ολοκληρωθεί αυτό το διάστημα των τριών ετών, να υπάρξει μια πραγματική μελέτη αντικτύπου για να δούμε αν υπάρχουν θετικέ και αρνητικέ συνέπειε για την Παππούα Νέα Γουινέα και τα νησιά Φίτζη και αν υπάρχουν θετικέ και αρνητικέ συνέπειε στον ευρωπαϊκό κλάδο, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια τελική λύση, να δούμε κατά πόσο μας ενδιαφέρει ή δεν μας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε το θέμα αυτό στο μέλλον. Αυτό ήθελα απλώς να σας πω. Ελπίζω να ήμουν σαφής και να σας έδωσα επαρκή στοιχεία ε, τα οποία υποστηρίζουν ε, τη θέση μου. Σε κάποιες περιπτώσεις η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου μάλλον αγνοεί κάποια πράγματα, τουλάχιστον την πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένες φορές ε, δεν βοηθάμε τρίτες χώρες και ε, σε αυτή την περίπτωση δεν βοηθάμε την Παππούα Νέα Γουινέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, είναι πολύ σοβαρό και θα πληρώσουμε ακριβά το τίμημα στο μέλλον. Αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση και να δώσω το λόγο στην κυρία Αντρέα Μπαρέα πολύ σύντομα, γιατί τρέχει και ο χρόνος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα που έγινε ε, με τις, τους κανόνες προέλευσης ε, στην Παπουανέου η νέα προκειμένου να υλοποιηθεί και η Ελία και τελικά δεν ε, έγινε και είχαμε ανάπτυξη από ορισμένε τρίτες χώρες ε, στο να κτίσουν εκεί τα εργοστία και να προβαίνουν σε μεταποίηση και κάνουν ντάμπιξ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ένα θέμα που πρέπει να το ξαναδούμε. Πολύ καλά τα είπατε, Πρόεδρε, στην περίπτωση αυτή. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε, όχι μόνο στην Επιτροπή Αλία γιατί αυτό ε, ουσιαστικά μπορεί να επηρεάσει και μελλοντικέ μας δράσεις, αλλά πρέπει να συνδυάσουμε τις δράσεις μας και θα πρέπει να έχουμε προσδιορισμό και της Επιτροπή ΣΥΝΤΑ, αλλά και του Επιτρόπου Εμπορίου, γιατί πρέπει να μας πούν ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι κανόνες και πρότυπα. Εγώ νομίζω ότι και γραπτές και προφορικές ερωτήσεις έχουν τεθεί στην Επιτροπή αλλά και στην Επιτροπή ΙΝΤΑ στην Επιτροπή Εμπορίου και εγώ θα ήθελα να ζητήσω μέγιστο συντονισμό και βάσει της ε, μελέτης της περιβαλλοντικής να δοθούν οι κατάλληλες εξηγήσει για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Κάποιος άλλος θα ήθελε το λόγο. Αλλιώς να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Καρσία Φερέρ. Μου είπαν ε, ότι η κυρία Γκαρσία Φερέρ ε, ήταν εδώ, αλλά τελικά δεν είναι. Ούτε ο κύριο Σιδεμπερέκ. Λοιπόν, τέλο πάντων, να πάρει το λόγο ο αρμόδιο από την Κομισιόν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το όνομά μου είναι Γιώχιμ Τσέλερ. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω αλλά θα δώσω τον ε, λόγο στην κυρία Γκαρσία Φερέρ και σε άλλους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ για να απαντήσουν. Αναφερθήκατε στους κανόνες προελεύσεως που προβλέπονται εις ε, την μεταβατική περίοδο. Θα ήθελα όμως να σας πω καταρχήν ότι υπάρχει μία συμφωνία την οποία έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007 με ε, χώρες της Καρεβικής και του Ειρηνικού για να υπάρχει μία συνέχιση στην πρόσβαση στην αγορά χωρίς προσωστώσει σύμφωνα με το προτιμησιακό σύστημα του Κοτονού που καλύπτεται από τον ΠΟΕ. Είναι μία προϋπόθεση για να υπάρχει αυτή η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, συμφωνία είναι προσωρινή αναφέρεται ιδίως σε εμπορεύματα και προσπαθούμε να συνάψουμε μία συνολική συμφωνία εφόλης της ύλη και με τις χώρες του Ειρηνικού έγινε ήδη μία τεχνική συζήτηση, θα υπάρξει μία δεύτερη και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε ε, στο τέλος να καταλήξουμε σε μία τέτοια ε, συμφωνία εταιρική σχέσης και ε, η ολοκληρωμένη αυτή συμφωνία θα μπορέσει να καλύψει πολλούς, πολλές περιοχές, θα έχει ένα πλήρες κεφάλαιο για την αλληλεία, για την αηφόρα διαχείριση των πόρων και ένα κεφάλαιο για τα κοινωνικά και εργασιακά θέματα και το περιβάλλον που δεν είχαν καλυφθεί στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρική σχέσης. Ο στόχος αυτής ε, της ε, συμφωνίας είναι ε, για τις για τις Φίτζι και τα PG να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά. Δεν υπάρχουν τελεσίδικες συμφωνίες με τις περιοχές αυτές, αλλά ελπίζουμε ότι οι Φίτζι θα μπορέσουν ε, σύντομα να εφαρμόσουν αυτή την ενδιάμεση συμφωνία εταιρική σχέσης. Όσον αφορά τους κανόνες προσέλευσης. Όπως εξήγησε η Πρόεδρος, προβλέπουν ε, για τα ε, ε, προϊόντα που χρησιμοποιούνται και δεν είναι αλλιευτικά και προβλέπονται ή στον κανονισμό αγοράς να μπορούν να συμπεριληφθούν ή στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης. Ο στόχος των κανόνων προελεύσεως ε, προτείνει να στηρίξει τις δυνατότητες λαμβάνοντας υπόψη την ειδική κατάσταση ε, της περιοχής όπου δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αλληλείας ή να προμηθευτεί προϊόντα τα οποία να συνάδουν με τους ε, συμπεφωνημένους κανόνες προελεύσεως που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε άλλες ενδιάμεσες συμφωνίες εταιρική σχέσης. Να τονίσουμε λοιπόν και να τονώσουμε την βιομηχανία και στην περιοχή PNG και εις τον ειρηνικό για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες αρχές οποιαδήποτε άλλη ενδιάμεση συμφωνία εταιρική σχέση απλούστατα λαμβάνοντας υπόψη για τον ειρηνικό τις ιδιάζουσες συνθήκες οι οποίες υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Ε, πρόκειται για έναν κανονισμό ο οποίος εφαρμόζεται από τις αρχές του 2008 μέχρι στιγμής ε, έχουμε περιορισμένες πληροφορίες ως προς τις επιπτώσεις των κανόνων προελεύσεως επί των πόρων επί της αναπτύξεως της αλληλείας στην περιοχή αυτή και όπως είπε η πρόοδος υπάρχει μία έκθεση που πρέπει να καταρτιστεί ε, για τις δραστηριότητες στο χώρο αυτό μέχρι του χρόνου το 2011 και ήδη έχουμε αρχίσει να ετοιμάζουμε την έκθεση αυτή για να είναι διαθέσιμη το 2011 και καλύπτουμε τα διάφορα θέματα όπου συγκεντρώνουμε αποδείξεις από, στις περιοχές που ανέφερε η Πρόεδρος. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία απόδειξη για αρνητικές επιπτώσεις των κανόνων προελεύσεως για την ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία ε, αλίας ή μεταποίησεως και οι εισαγωγές ε, αντιπροσωπεύουν μόνο 3% των συνολικών εισαγωγών τόνου παραδείγματος χάνει και συναδελφός μου θα σας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άρα αυτή τη στιγμή ε, η συμμετοχή αυτών των ε, ενδιαμέσων συμφωνιών εταιρική σχέση σχετικά με τον τόνο είναι αμεληταία και δεν θα μπορούσε να έχει σημαντική επίπτωση στην αλληλεία στην Ευρώπη και αυτό ήταν ένας από τους κανόνες που λήφθηκαν υπόψη όταν ε, καταρτήσαμε τους κανόνες προελεύσεως για τον ε, ειρηνικό. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι όσον αφορά την δυνητική ανάπτυξη των περιοχών αυτών, όντως ε, υπάρχουν ε, επιταγές ε, που ρυθμίζουν την παράνομη αλληλεία άπαξ και εφαρμοστούν οι συμφωνίες και θα πρέπει να εφαρμοστούν επίσης και οι κανόνες για τις υγειονομικές προδιαγραφές που είναι η βάση της, των προϋποθέσεων εξαγωγής αλληλευτικών προϊόντων προς την Ευρώπη όσον αφορά το, την αλία υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις αλλά δεν θέλω τώρα να επισέλθω σε λεπτομέρειες και δεν έχουμε κάποια, ε, κάποιο στοιχείο που να μας δείχνει ότι υπήρξε σημαντική επίπτωση των ε, ενδιαμέσων συμφωνιών εταιρικής σχέσης ε, στην ε, Ευρώπη ή ότι επηρεάζουν την βιομηχανία. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο λίγες πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις των επενδύσεων σε ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης. Υπάρχουν δηλαδή μόνο δύο περιπτώσεις που μπορούν και έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε ε, κονσερβοποιίες στην περιοχή για εξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δουλειές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είναι ιδίως για γυναίκες και για τους ντόπιου στις κονσερβοποιίες αυτές, αλλά είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε λεπτομερώς εις την μελέτη κανόνων προελεύσεως που καταρτίζουν για τον επόμενο χρόνο. Και υπάρχει στο παράρτημα μία διάταξη που προβλέπει την αναθεώρηση των κανόνων προελεύσεων βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής για την εφαρμογή των κανόνων προελεύσεως. Βέβαια έχουν περάσει μόνο δυόμιση χρόνια, δεν έχουμε ε, μία αρνητική απόδοση απόδειξη της επιρροής στα βιώσιμα αποθέματα στον ειρηνικό και με αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε την ποσότητα των αλλιευμάτων στον ειρηνικό που θα ληφθούν υπόψη στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρική σχέσης. Το θέμα το, της διαχειρίσεως των πόρων στον ειρηνικό, των αλληλευτικών ε, πόρων στον ειρηνικό, πρέπει να ληφθεί υπόψη ή στις εξετάσεις από διάφορους εμπλεκόμενους για να περιοριστεί η πρόσβαση, να, χρειάζονται, ε, να χρειάζεται χορήγηση ε, άδεια στα πρώτα πλοία τα οποία προτίθενται να να ε, ψαρέψουν στην περιοχή για να στηρίξουμε την ε, αηφόρο διαχείριση ε, πόρων ή στον ειρηνικό και μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει κάποια αρνητική επίπτωση ή σημαντική αύξηση ή στις τις ε, αλλιευτικές δραστηριότητες στον Ειρηνικό σχετικά με την ε, ονομασία προελεύσεως. Δεν υπάρχει δηλαδή ε, κάποια αντική επίπτωση από τις ενδιάμεσες συμφωνίες εταιρικής σχέσεως και τις τις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Πρόεδρε, προσπάθησα να ε, απαντήσω σε ορισμένα θέματα και αν επιτρέπετε οι συνάδελφοί μου μπορούν να προσφέρουν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο στην περιοχή. Εντάξει, αν κάτι πολύ ε, σύντομο έχετε να προσθέσετε, εντάξει, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο γιατί πρέπει να διακόψουμε για το γεύμα. Έχουμε και τα ωράρια των δερμηνέων. Εγώ όμω ε, θέλω να πω το εξή. Αν εσεί ήδη στο στάδιο αυτό κάνετε μια έκθεση αξιολόγηση για να δείτε αν λειτουργεί όχι η παρέκκληση και όταν ξέρετε ότι δεν εφαρμόζεται στο φίτσι και όταν ε, αρχίζει να ε, αναπτύσσεται η μεγάλη ζώνη στο Ματούν. και εγώ βλέπω ότι ε, σε δύο χρόνια η πρόβλεψη είναι στους 400.000 τόνους. Τώρα βλέπετε ότι ήδη μειώνεται ο αντίκτυπος, αλλά εγώ θα ήθελα να δω ποιος είναι ο αντίκτυπος μέσα σε δύο χρόνια. Τώρα αυτή η αξιολόγηση σε τίποτα δεν χρησιμεύει, γιατί δεν έχουμε τις ποσότητες που θα μπορούσαν να παραχθούν ή που προτείνετε να παραχθούν. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, λέτε ότι δεν είχατε καμία ενημέρωση για την αλία απλά παράνομη λαθρέα και ανάρχη αλεία. Όμω, ε, κοιτάξτε, δεν θα σα στείλουν αυτοί που αλλιεύουν ε, παράνομα αυτέ τι πληροφορίε. Χρειάζεται χρόνο. Και ε, επίση πρέπει να δούμε τι γίνεται όταν μιλάμε για ένα τέτοιο είδου αλεία. Εσεί Μιλάτε τώρα για ένα θέμα το οποίο θα δούμε τον αντίκτυπο σε δύο χρόνια. Έτσι λοιπόν αυτό που θα κάνετε τώρα θα είναι τα ίδια που κάνατε πριν. Αυτό δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο γιατί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε ποιε είναι οι προβλέψεις που κάνουν οι ίδιοι για τα επόμενα δύο χρόνια. Και εγώ χρησιμοποίησα τι προβλέψει. Τώρα σήμερα φυσικά και δεν υπάρχει κανένα αντίκτυπο. Πώ θα έχει αντίκτυπο σήμερα. Όμως γνωρίζοντας ε, το τι συμβαίνει στην ε, Τιλανδία, γνωρίζοντας στην Ταϊλάνδη τα σχετικά στοιχεία των Φιλιππινών λιγότερο, εγώ σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και μου δίνεται η εντύπωση ότι ε, το ίδιο γίνεται και εκεί με αυτά τα κατόφλια που έχετε καθορίσει. Εγώ για την Ταϊλάνδη το ξέρω από πρώτο χέρι και νομίζω ότι τα εργοστάσια που έχουμε εκεί είναι τελανδέζικα εργοστάσια. Κοιτάξτε, πολύ αμφιβάλλω ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα στην περίπτωση αυτή. Εσείς ξέρετε πολλά από εμπόριο, ξέρω πολλά από αλία. Αυτή είναι η διαφορά που έχουμε μεταξύ μας. Και αυτό είναι και το πρόβλημα. Λοιπόν, όπως και να έχει, ξέρετε, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και για το έργο σας και σας ζητώ να σημειώσετε το τι λέμε εδώ και να το διαβάσετε στη γάμα δέλτα μάρε. Ε, ίσως θα ήταν ε, καλύτερο ε, στο μέλλον να προσπαθήσουμε καλύτερα να συνοηθούμε μεταξύ των δεμένων εμπορίου και ελίου. Βέβαια δύσκολο σήμερα. Τώρα, για το θέμα της χιλής, καθώς έχει περάσει η ώρα, θα το δούμε για το απόγευμα μετά από το σημείο 10. Έτσι λοιπόν διακόπτουμε τώρα μέχρι τις 3 και θα δούμε το σημείο που μας έμεινε.